Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me to open today's afternoon meeting of Regi. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Οι συνάδελφοι που είναι απόντες ελπίζω να έρθουν σύντομα. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι με χαρά ε, υποδέχομαι τον αρμόδιο υπουργό από τη Ρουμανία, την κυρία Πλάμπ δηλαδή. Είναι προεδρεύουσα από την 1η Ιανουαρίου και με χαρά σήμερα θα ακούσουμε τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας και θα συζητήσουμε και τις ε, περιφερειακές πολιτικές με την Υπουργό κυρία Πλούμπ. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Υπουργό να παρουσιάσει τις θέσεις της και μετά τα μέλη της Επιτροπής για ερωτήσεις, σχόλια και θα ανταπαντήσει η Υπουργός Πλάμπ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι μαζί σας ξανά σήμερα για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ρωμανικής Προεδρίας Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα την οποία μας δίδεται το πρόγραμμα της Ρουμανικής Προεδρίας έχει σαν βασικό στόχο να συνεισφέρει στην επιτυχία της πολιτικής ατζέντα του πολιτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένα θέματα όπως η πολιτική συνοχής. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουμε στα πλαίσια της εναλλασσόμενης Προεδρίας είναι μια δύσκολη θα έλεγα περίοδος, υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες οι οποίες αφορούν και στην καθημερινότητα των πολιτών και στις ε, κυβερνητικές εξελίξεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε με συνολικό τρόπο να ε, φέρουμε εις πέρα στην αποστολή μας. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι και κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών και συνεπώς θέματα όπως το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Αλλά είμαστε και φιλόδοξοι, θα προσπαθήσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, σημειώνοντας πρόοδο σε ορισμένα σημαντικά θέματα Εμείς θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε αντικειμενικά ως διευκολυντές και ενδιάμεση για να προωθήσουμε τις διαφορετικές θέσεις. Η ε, Προεδρία της Ρωμανίας θα είναι μια Προεδρία των πολιτών. Η βασική μας στόχη είναι να προωθήσουμε και νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών και να συνεισφέρουμε σε μία, για μία μάλλον ένωση η οποία να είναι πιο δημοκρατική και πιο κοντά στους πολίτες. Ελπίζουμε η συνάντηση κορυφής του ΣΥΜΠΙΟΥ στις 9 Μαΐου να είναι μια σημαντική φάση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση νομίζω ότι θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε μια πληρέστερη, συνεκτικότερη και δημοκρατικότερη ενωτική Ευρώπη. Το μόντο, το βασικό μας σύνθημα αν θέλετε, αντικατοπτρίζει τις ανάγκες τις οποίες έχουμε για ενότητα και συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη όπως επίσης και την ανάγκη για περισσότερη οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή όπως προβλέπουν οι συνθήκες. Ε, βλέπετε εδώ το σήμα μας, ένα ιστορικό πρόσωπο, ε, είναι κάτι το οποίο μεταφέρει θα έλεγα την ε, ισχυρή βούλησή μας να πετύχουμε. Η στόχοι μας σε νομοθετικό και σε μη νομοθετικό πεδίο ε, ανήκουν σε τέσσερα, θα έλεγα, σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς. Συνοχή, παγκοσμιοποίηση, κοινέ αξίες, εξωτερική πολιτική. Ε, θα συγκεντρωθώ περισσότερο σήμερα εδώ στον πρώτο πυλώνα, γιατί συνδυάζει νομοθετικά θέματα με τα οποία έχετε ασχοληθεί. Η σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια περίπτωση από όπου όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές συνεισφέρουν στη μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών διαφορών. Η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζεται φυσικά άμεσα από τις ε, δυνατότητες σύγκλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς η συνοχή, η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι οι βασικές προτεραιότητες για τη Ρουμανία. Το νομοθετικό πακέτο για την πολιτική συνοχή αποτελεί ένα σημαντικό θα έλεγα στάδιο στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Εμείς εδώ ε, θα εκφραστούμε θετικά για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα σχετικά με τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους, την βελτίωση της ευελιξίας και της αναλογικότητας. Αυτά θα έλεγα δείχνουν τις φιλοδοξίες που έχουν και τα δύο νομοθετικά όργανα να απλοποιήσουν την πολιτική συνοχή, να την καταστήσουν αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη για τους δικαιούχους στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής μας ε, θα έλεγα εντολής. Εμείς θα συνεχίσουμε και σε κάποιους τομείς τους οποίους ξεκινήσαμε κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας και θα εξετάσουμε το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων της συνοχής ιδιαίτερα σχετικά με τον κανονισμό πλαίσιο. Βασικός στόχος της Ρουμανικής Προεδρίας είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με δυναμικό τρόπο, διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντικές ε, ε, αποφάσεις και σε σημαντικά βήματα προόδου, να προετοιμάσουμε τον τριγωνικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε το νομοθετικό πακέτο να προετοιμαστεί έγκαιρα και να θέσει τα θεμέλια για μια επιτυχή πολιτική για την επόμενη περίοδο η Ρουμανική Προεδρία έχει σαν βασικό στόχο να λειτουργήσει αντικειμενικά σχετικά με τον κανονισμό και τα θεματολογικά μπλοκ του κανονισμού αυτού, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας και των συζητήσεων για το πολιετές δημοσιονομικό. Θα συνεχίσουμε εμείς τις διαπραγματεύσεις για τα υπόλοιπα έξι θέματα οι ομάδες θεμάτων, δηλαδή πλαίσιο επιδόσεων, οικονομική στήριξη από τα ταμεία, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση, υποπτία, αξιολόγηση, επικοινωνία, καλύτερη ορισμοί και φυσικά το ίδιο το δημοσιονομικό πλαίσιο. Για το ERDF και για τα ταμεία συνοχής, η Ρουμανική Προεδρία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις επί τη βάση της προόδου που έχει επιτελεστεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης Προεδρίας, της Αυστριακής, έτσι ώστε να καταλήξουμε σήμερα σε κοινέ θέσει. Το ίδιο επίσης και για το μπλοκ 2, για το Interreg. Δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος μέχρι τώρα για να μπορέσουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εντολή για το Συμβούλιο, από το Συμβούλιο. Οι συζητήσεις όμως ξεκίνησαν αυτό το μήνα σε τεχνικό επίπεδο. Θα σημειωθεί ελπίζω πρόοδος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον μήνα Ιούνιο. Εμείς ε, θα επωφεληθούμε από τα βήματα των διοργανικών συζητήσεων και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε τεχνικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή οι δύο συνομοθέτες προετοιμάσουν τις εντολές τους το Συμβούλιο έχει μια εντολή διαπραγμάτευσης για τον μπλοκ υπαρίθμ 1, προγραμματισμός και στρατηγική, PIPS, όπως επίσης και διαχειριστικές προβλέψεις. Μια συμφωνία στην οποία είχαν καταλήξει γι' αυτά κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας. Συνεπώς η Ρουμανική Προεδρία θα έχει σαν στόχο να υπάρξει μια ειδική συνάντηση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την Πολιτική Συνοχή, στα πλαίσια του οποίου οι Υπουργοί θα επικυρώσουν την πρόοδο η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου. Στις υπόλοιπες πολιτικές συνοχής απαιτείται ένα καλύτερο πλαίσιο συνεργασίας, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποια επιμέρους κοινά θέματα στα πλαίσια των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι θα ότι η Ρουμανική Προεδρία και το Συμβούλιο θα μας οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα. Συνειδητοποιούμε ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν θα τα πετύχουμε αν δεν μας έχουν υποστηρίξει όλες οι χώρες μέλη. Εμείς λοιπόν υπολογίζουμε και στη δική σας υποστήριξη ιδιαίτερα της δικής σας κοινοβουλευτικής επιτροπής, είναι απαραίτητη για να πετύχουμε κι εμείς. Τα πιο σημαντικά θα έλεγα σημεία για την πολιτική συνοχή, τα οποία σκοπεύουμε να οργανώσουμε εμείς κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας, θα είναι η ανεπίσημη ε, συνάντηση Υπουργών για τη Συνοχή στις 11 και στις 12 του μηνός Απριλίου ανεπίσημη επίσης συνάντηση για τον Τέρμπαν στις 13 και στις 14 Ιουνίου, όπως επίσης και η συνάντηση κορυφής της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία θα οργανωθεί στις 13, 14 και 15 Μαρτίου. Θα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι φυσικά να σας ζητήσουμε να είσαστε παρόντες κατά τη διάρκεια αυτών των τριών συναντήσεων. Να σημειώσω επίσης ότι η Προεδρία μας είναι απόλυτα δεκτική. Θέλουμε να έχουμε έναν δίκαιο διάλογο μαζί σας. Θα σας ακούσουμε. Θα ακούσουμε φυσικά και τα κράτη-μέλη και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να προχωρήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα και στο νομοθετικό πακέτο για την πολιτική συνοχή που έχει τόσο μεγάλη σημασία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις μάχες τις οποίες δώσατε μέχρι τώρα. Έχετε πετύχει πολλά στην προώθηση της πολιτικής συνοχής. Είναι η πιο σημαντική θα έλεγα ε, πολιτική σε επίπεδο επενδυτικό για το μέλλον της Ένωσης. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε επί τη βάση της μέχρι τώρα συνεργασίας μας. Είπαμε δίκαιος διάλογος, ισότιμος διάλογος. Έτσι θα πετύχουμε να οικοδομήσουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ισχυρό προς όφελος του συνόλου των Ευρωπαίων πολιτών. Έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε επίσης σε τους στόχους μας στην αηφόρο ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα, προς όφελος ε, του συνόλου επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά των Ευρωπαίων πολιτών. Είμαι πεπισμένη ότι θα το πετύχουμε. Είμαι επίσης πεπισμένη ότι η Ρουμανία ως προεδρεύουσα θα λειτουργήσει συλλογικά και θα προασπιστούμε την πολιτική συνοχής. Θα λάβουμε υπόψη μας τη στενή σχέση της πολιτικής συνοχής με το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό και είμαι σίγουρη ότι θα καταλήξουμε σε σωστά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε τις απόψεις σας και χαίρομαι που ξαναγύρισα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για αυτά τα οποία έχετε κάνει, για αυτά τα οποία κάνετε και θα σας ακούσω με προσοχή και ελπίζω να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you, Minister. And, uh, now... Ευχαριστώ, Υπουργέ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη και στους προσκεκλημένους μας. Συνήθως ήρθατε να ξεκινάμε με τους συντονιστές. Έχουμε τρεις στην συνεδρίαση σήμερα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους συντονιστές και μετά θα, θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μέλη. κυρία Κρέλ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, χαίρομαι ιδιαίτερως ε, που είστε εδώ και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα λίγα λεπτά. Αλλά σήμερα έχουμε την... από την ε, περιφερειά μου στη Γερμανία και ήθελα να ακούσουν και αυτοί πώς πήγε η ψηφοφορία σε ό,τι αφορά τον ε, κανονισμό της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Γι' αυτό και καθυστέρησα λίγο. Καταρχάς, χαίρομαι λοιπόν που η Ρουμανική Προεδρία δίνει τόσο σημαντική, τόσο μεγάλη προτεραιότητα στην πολιτική συνοχή. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μια πολιτική ένδειξη σημαντική για τα κράτη-μέλη. Το θέμα της αλληλεγγύης και των σχετικών επενδύσεων στην Ευρώπη πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Και ελπίζω αυτό να δημιουργήσει με τη σειρά του και παραπάνω εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσουμε λοιπόν έτσι ένα μήνυμα ότι οι επενδύσεις ε, σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχιστούν. Και με την ε, απαραίτητη δέσμευση. Σήμερα το πρωί θα τα ακούσατε. Ψηφίσαμε σε ό,τι αφορά το γενικό κανονισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι ε, συμμετείχαν και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα που πετύχαμε είναι πολύ καλό και ελπίζω ότι με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου θα λάβουμε και την εντολή να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή και να ξεκινήσουν ε, οι διαπραγματεύσεις με την Προεδρία. Αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι και είναι ευθύνη των ερετών ε, βουλευτών να κάνουν τη δουλειά τους ε, σωστά πρωτού ξεκινήσουμε τον προεκλογικό αγώνα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε τις ευθύνες μας ε, για να αντιπραγματευτούμε στο βαθμό του δυνατού την ε, πολιτική συνοχή. Χαίρομαι που θέσατε το θέμα της διαχείρισης ε, και του management. Αν καταφέρουμε να περάσουμε και άλλα τέτοια κομμάτια, το Κοινοβούλιο σίγουρα θα είναι δεθμένο να τα πετύχει όλα αυτά. Και ελπίζω τον Απρίλιο να έχουμε ολοκληρώσει ήδη κάποιες ενότητες του κανονισμού. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι ωφέλιμο όχι μόνο για τις εργασίες του Κοινοβουλίου, αλλά θα αποτελέσει και ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης ε, στους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν καταβάλουμε λοιπόν κάθε προσπάθεια για να συνεχιστούν αυτές οι δυνατότητες επένδυσης. Ακόμα και αν δεν θα είναι η Προεδρία σας αυτή που θα δημιουργήσει το οικονομικό πλαίσιο, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να προχωρήσουν τα θέματα αυτά. Και να ξεκινήσει ο προγραμματισμός αυτός. Σήμερα λοιπόν ψηφίσαμε το Γενικό Κανονισμό στην ε, Επιτροπή αλλά στον Interreg θα πάρουν το λόγο φαντάζομαι και οι σκιώδες συζήτητες για να μιλήσουν. Προγραμματίζονται λοιπόν ε, οι πρώτε συναντήσει. Ελπίζω λοιπόν και με το Ταμείο Συνοχή να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και το αργότερο να περάσει το θέμα αυτό στην Ολομέλεια το Μάρτιο για να ξεκινήσει και ο τρομερή διάλογο. Αυτό πιστεύω ότι ανταποκρίνεται και στις ευθύνε που έχουμε έναντι των Δήμων και των κοινοτήτων, αλλά έναντι και των πολιτών. Ελπίζω να έχετε την ευκαιρία να προχωρήσετε τα θέματα αυτά, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό ως μήνυμα από πλευρά της Προεδρίας. Δεν είχα συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι πρόκειται για την πρώτη Ρουμανική Προεδρία και το μόνο που έχω να πω είναι ότι σας ευχόμαι κάθε επιτυχία. Είναι πάρα πολύ σύντομη φυσικά το χρονικό διάστημα σε ό,τι φορά και τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σταθεί με επιτυχία η Προεδρία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λέει πρόεδρος. Η κυρία Μασίτσου. Ευχαριστώ, πρόεδρε, κυρία Τόμασίτσου. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ στην ε, Επιτροπή μας. Χαίρομαι ιδιαίτερος που η Ρουμανία προεδρεύει στο Υπουργικό Συμβουλίο. Η Κροατία θα ξεκινήσει και θα έχει την πρώτη προεδρία το 2020. Πολλά νομίζω ότι μπορούμε να ενταχθούμε από εσά. Σα εύχομαι κάθε επιτυχία, γιατί έχετε και πολλού τρομερεί διαλόγους σε ό,τι αφορά τα θέματα τη περιφερειακής ανάπτυξη. Ελπίζω να καταφέρετε να ολοκληρώσετε του πιο πολλού εξ αυτών. Δυστυχώ έχουμε και εκλογέ μπροστά μα. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μα αυτό. Ελπίζω να έχετε ε, μεγάλη επιτυχία και να μας ε, δείξετε ότι οι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη μπορούν και αυτέ να κάνουν πολύ καλή δουλειά και ότι δεν ε, του ε, πήγε να φέρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά λαμβάνουν τι αποφάσει του ε, υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και καλώ ορίσατε, κύριε Υπουργέ. στην Επιτροπή μας από πλευρά της ε, ομάδας των φιλελευθέρων. Όπως σας είπα, όπως είπατε μάλλον, η πολιτική συνοχή είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες ε, της Προεδρίας σας. Στα αγγλικά όμως, ξέρετε τι λέμε, ότι τελικά εκ των υστέρων θα φανεί, θα προκύψει. Και έχω να πω το εξή. Δεν υπάρχουν πολλέ λεπτομέρειε στο πρόγραμμα. Γιατί? Και για να το πάω και παραπέρα. Αναφέρθηκε το Interreg και το άλλα ζητήματα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ε, Διασυναριακών Μετακινήσεων κτλ. Ρωτώ λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν ακόμα προτεραιότητα για την Προεδρία σας ε, και ποια είναι τα βασικά εμπόδια τα οποία καλείστε να αντιμετωπίσετε, να αντιμετωπίσετε στο Συμβουλίο. Τι θα κάνετε επίσης για να υπερπηδήσετε τα εμπόδια αυτά προκειμένου να ξεκινήσουν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις. δεν σχετίζεται αυτό με το πουδουπού, καθότι δεν υπάρχει η διάσταση αυτή, η χρηματοοικονομική. Από το Βουκουρέστι, λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να βρείτε μια γενική προσέγγιση για τα θέματα αυτά, σε ό,τι αφορά την όλη διαδικασία της διαπραγματεύσης. Ω Επιτροπή έχουμε εκφράσει την ανησυχία μα ότι πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τον κανονισμό για τις γενικέ διατάξεις μπαίνουν στο παιδεία διαπραγμάτευση. Δηλαδή, το Συμβούλιο πολύ αργά, πολύ απλά θέλει πρώτα να συμφωνήσει και μετά να έρθει να μας τα παρουσιάσει όλα αυτά. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεν σέβεται αυτό τη εξουσία και τι αρμοδιότητε του συνομοθέτη. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η δική σα τοποθέτηση και τι θα κάνετε για να μα επιτρέψετε να διαπραγματευτούμε και πέρα από τα σημεία αυτά που αναφέρατε στην παρουσίασή σας. Και τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια τοποθέτηση για τον κανονισμό για την προστασία του ευρωπαϊκού προπολογισμού σε περίπτωση γενικευμένων ζητημάτων σε ό,τι αφορά το, τα θέματα κράτους δικαίου τα κράτη-μέλη. Ο μηχανισμός κράτους δικαίου, όπως αποκαλείται. Πολύ σημαντικός φάκελος για μένα και θεωρώ ότι πραγματικά χρειάζεται για να είναι επιτυχές το πολιτισμό στο πλαίσιο μετά το 2020. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου και αυτό ενδεχομένω να επηρεάσει τα συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ και η δική σα χώρα, η Ρουμανία, συγκαταλέγεται στι χώρε αυτέ. Υπάρχουν σοβαρέ αμφιβολίε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου. Ερωτώ λοιπόν, τι θα κάνετε για να προωθήσετε τα θέματα αυτά. Υπάρχει δυνατότητα να πετύχετε ε, γενική πρόοδο υπό την Προεδρία σας και τι προσπάθειες θα καταβάλλετε για να σημειωθεί πρόοδο στο θέμα αυτό. Σχετίζεται αυτό άλλωστε και με τη χρηματοδότηση διαφόρων δράσεων μεταξύ των οποίων και η πολιτική συνοχή προφανώ. Να σας ευχηθώ λοιπόν κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας και φαντάζομαι ότι είσαστε συνεπαρμένοι στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα να σας ε, διαβεβαιήσω ότι και από δική μα πλευρά, από πλευρά τη ομάδα των φιλελευθέρων, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να στεφτεί η Προεδρία σα με επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Επόμενο μελετή, ο κύριο Μπούντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, καλώ ορίσατε στο Κοινοβούλιο και να σα ευχηθώ και εγώ κάθε επιτυχία για την Προεδρία σα είναι σημαντικό, γιατί η δική σας επιτυχία θα σημαίνει επιτυχία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύρια Υπουργέ, κάναμε συζητήσει και με δημάρχους, όχι μόνο στη Ρουμανία, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη και καταγγέλουν πόσο δυσκίνητη είναι η διαδικασία σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την κινητοποίηση πόρων. Και πολύ συχνά διαπιστώνουμε ότι οι κανόνε του παιχνιδιού αλλάζουν. Αλλάζουν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Και στη Ρουμανία λοιπόν άλλαξαν πρόσφατα οι αρμοδιότητες των αρμόδιων αρχών. Αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά τη χρήση των μέσων αυτών. Ερωτώ λοιπόν, Τι έχετε να πείτε για την ανάγκη πραγματική απλοποίηση των διαδικασιών. Και άλλη μια ερώτηση από πλευρά των Βρυξελών. Τα κράτη-μέλη. Μάλλον επιβάλλονται στα κράτη-μέλη δύο-τρία επίπεδα διατάξεων, αλλά και στο τοπικό επίπεδο επιδεινώνεται η κατάσταση και περιπλέκονται οι προδιαγραφέ. Αυτό το έχουν καταγγείλει πολλά κράτη-μέλη. Ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχουν διάφορα έργα τα οποία διεξαγάγονται σε εθνικό, κεντρικό επίπεδο, ενώ το τοπικό επίπεδο ε, δηλώνει ότι θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα προγράμματα αυτά και σε κάποιε περιπτώσει δεν ήταν εκεί η συνεργασία μεταξύ τοπικού και κεντρικού επίπεδου. Θα μπορούσατε μήπω να προωθήσετε την διεξαγωγή όλων των προγραμμάτων αυτών και την αρμοδιότητα σε τοπικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την πραγματοποίηση ευρωπαϊκών έργων. Μία τελευταία τώρα ερώτηση. Και σε ό,τι αφορά τι κοινωτικέ αρχέ, Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μία δομή για την υποβολή ετοιμάτων χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Να υπάρχει δηλαδή τοπική, τοπικός μηχανισμός στο τοπικό επίπεδο για την ανάληψη πρωτοβουλειών και για την υποβολή ετοιμάτων χρηματοδότησης. Άλλη μία παρατήρηση. Μιλήσατε για μια ισχυρή πολιτική συνοχή, αλλά δεν βάλατε ως προτεραιότητα το ίδιο κεφάλαιο για τη σημερινή ψηφοφορία. Το θέμα της μακροοικονομικής ρεσιμότητας, πώς ε, τοποθετείται έναντι αυτού η Ρουμανική Προεδρία και σε ό,τι αφορά τη συγχρηματοδότηση. Πείτε μας ποια είναι η στάση της Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ο επόμενος μιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως εισηγητής για το Ιντερεκ, θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να παρουσιάσω και εγώ τις δικές μου ερωτήσεις και αξιώσεις προς την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Είμαι εισηγητής άλλωστε για ένα θέμα προστασίας των καταναλωτών. Έχουμε σήμερα το βράδυ μάλιστα ένα σχετικό τριμερή διάλογο και τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά γρήγορα. Έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο σε ό,τι αφορά την Ρωμανική Προεδρία θα ήθελα να πω θα ήθελα να τα έχουμε αυτή την επιτυχία και στις, στα θέματα της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το 2017 μας είπαν ότι αν αναλάβουμε το θέμα αυτό έπρεπε να φροντίσουμε να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μέχρι το τέλη του επόμενου έτους και να έχει ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο. Γιατί στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τρεμερεί διαλόγου με τη Ρουμανική Προεδρία προκειμένου να πετύχουμε όσο μεγαλύτερη συμφωνία γίνεται πριν από τι ευρωεκλογέ υπό τη Ρουμανική Προεδρία. Αυτό λοιπόν και το κάναμε από πλευρά ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά ταμεία, το Κοινοβούλιο εργάστηκε ταχύτατα στον τομέα του Interreg. Είχαμε μια μόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα καταφέραμε λοιπόν να το πετύχουμε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Με μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίστηκε το θέμα αυτό. Και ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από καμία πολιτική ομάδα. Όλοι πιστεύουμε ότι το Interreg θα πρέπει να συνεχιστεί ως εργαλείο, ω μηχανισμό Είναι καλό εργαλείο. Έχουν νόημα αυτά τα έργα και προωθείται η διασυνοριακή συνεργασία η οποία είναι πιο σημαντική από ποτέ. Όλα αυτά τα λέω για να σας πω ότι είμαστε πανέτοιμοι να διαπραγματευτούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή η γενική προσέγγιση θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Αυτό θεωρώ Ε, σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα αυτού του δύο-τρει μήνε, τέσσερι μήνε. Ε, γιατί θα καταρτίζει την γενική προσέγγιση του Συμβουλίου. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί θα μπορούσαμε να καθορίσουμε σε μεγάλο βαθμό το κοινό αυτό κείμενο. Και αν ε, η Ρουμανική Προεδρία θεωρεί ότι τα αδερφατικά ταμεία είναι σημαντικό θέμα και ότι αξίζει τον κόμπο από πολιτική άποψη να το υποστηρίξει, εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει πολλά σημαντικά αποτελέσματα. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, κάτι τέτοιο δεν ε, πρόκειται να γίνει και θα ήθελα να σας παρακαλέσω το εξή. Ίσως θα μπορούσατε να προσαρμόσαστε την ατζέντα σας, προκειμένου και ο φάκελο αυτός να μπει σε φάση διαπραγμάτευση, γιατί ουσιαστικά ό,τι είναι... Ήταν να γίνει, έχει γίνει. Δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει η επόμενη, το επόμενο κοινοβούλιο, τι θα γίνει. Είναι ευκαιρία λοιπόν να προωθήσουμε το κείμενο αυτό, το οποίο άλλωστε το υποστηρίζει και το υποστηρίζουν και τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν μια έκκληση προς πλευρά σας. Ίσως θα μπορούσαμε στο θέμα αυτό, όπως και στο CPR, ίσως θα μπορούσατε λοιπόν να ολοκληρώσετε πολύ γρηγορότερα την γενική αυτή προσέγγιση και να μην χάσουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε τη διαπραγματεύση το θέμα αυτό πριν από τις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ κύριο Νοβάνκοφ. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να συγχαρώ την Υπουργό για θέματα περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχής, ιδιαίτερα για τον ενεργό ρόλο που έχει τραγματίσει ω τώρα και μετά από τι σημερινέ ψηφοφορίε θεωρώ ότι κάναμε ένα μεγάλο βήμα προ τα εμπρό και μεγάλη πλειοψηφία ε, εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή μα ε, θα συνεχίσει να εργάζεται στο ΣΥΠΙΑ. Και φυσικά, ω συνεισηγητή, θα ήθελα να μα πείτε ποια είναι η απόψή σα για τα πιο πολλά σημαντικά αυτά θέματα, αλλά κυρίω ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Και αυτό γιατί εδώ... μια και εμεί είμαστε υπεύθυνοι να προωθήσουμε τους φακέλους αυτούς. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ή μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον. Η ευθύνη, όλοι συμφωνούμε, είναι πολύ πιο ευρεία. Δεν αρκεί να μιλησουμε με καποιον η ευθυνη ολοι συμφωνουμε ειναι πολυ πιο ευρια δεν αρκει να ολοκληρωσουμε τη δικασία στο Κοινοβούλιο. Ουσιαστικά έχουμε ευθύνη εναντί κάθε δικαιούχου, κάθε μικρομεσαίας επιχειρήσεις, επιχειρήσης, ε, κάθε πολίτη εργατή των δημάρχων, των δήμων, των κοινοτήτων. Όλοι τους ζητούν, απαιτούν απαντήσεις. Ποιες θα είναι οι προδιαγραφές, ποιοι θα είναι οι κανόνες από Ιανουάριο του 2021, ποια θα είναι τα κριτήρια, οι προδιαγραφές, ε, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικό λοιπόν να μας πείτε ε, εδώ και τώρα σήμερα στην Επιτροπή μας. Είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τις διαπραγματεύσει και ποιο χρονοδιάγραμμα θεωρείτε ότι θα ήταν ρεαλιστικό και σωστό. Δεδομένου ότι έχουμε ψηφοφορία στις 14 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζωάννα, έχει το λόγο. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ. Νομίζω ότι η παρουσία σας ήταν εξαιρετικά χρήσιμη στα νέα καθήκοντα που έχετε αναλάβει στη Ρουμανική Προεδρία. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και εμείς που εκπροσωπούμε τη Ρουμανία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας είμαστε ευγνώμονες για αυτή. Είναι ατού η εμπειρία σας για τη δική μας Επιτροπή για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και ως μέλος αυτής της Επιτροπής θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να υπογραμμίσω το γεγονός ότι έχουμε εξαιρετική συνεργασία ε, για όλους τους φακέλους που συζητούνται στην Επιτροπή μας. Παρακολουθήσατε εκ του Συνήκη τις εξελίξεις για τις υποθέσεις που μας αφορούν και που μας ενδιαφέρουν στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και μας βοηθήσατε ε, τότε τη στιγμή που το χρειαστήκαμε και όχι μόνο μία φορά. Επομένως, κυρία Υπουργέ, κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η Ρουμανική Προεδρία θεωρεί την πολιτική συνοχή ως απόλυτη προτεραιότητα, γιατί αυτό πράγματι στέκεται στο ύψος των προσδοκιών του Ευρωπαίου πολίτη και του Ρουμάνου πολίτη. Οι Ρουμάνοι πολίτες, όπως και οι λοιποί Ευρωπαίοι, έχουν ανάγκη να ε, βλέπουν επενδύσεις να γίνονται και μάλιστα στο τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε επενδύσεις και περισσότερη σύγκληση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των λοιπών πολιτικών όπως είναι η γεωργική πολιτική. Πρέπει να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της ε, ερήμωσης της ε, υπαίθρου. Δεν πρέπει να κρύψουμε αυτό το φαινόμενο Δυστυχώ, Είμαι μέλο και στην Επιτροπή Γεωργίας που συζητούνται αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνεργαστούν οι δύο επιτροπέ. Η έκθεση που ψηφίσαμε σήμερα λοιπόν ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Και εγώ η ίδια ήμουν εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση τη επιτροπή γεωργία σε σχέση με τον κανονισμό για τι κοινέ γενικέ διατάξει για το, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα λοιπά ταμεία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και το καθεξής εγώ λοιπόν μια ερώτηση να σας θέσω. Ποια είναι η θέση της Ρουμανικής Προεδρίας ως προς την έκθεση η οποία θα ψηφιστεί πριν από τις ευρωεκλογές στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, σας συγχαίρω για την παρουσία σας εδώ και για το έργο σας, για τα καθήκοντα που έχετε αναλάβει. Έχουμε την εντύπωση ότι η Ρουμανική Προεδρία θα διαρκέσει 3,5 μήνες αντί για τους 6 συνήθεις μήνες, ίσως λόγω των ευρωεκλογών. Είναι μια Προεδρία η οποία λαμβάνει χώρα ακριβώς πριν από τις ευρωεκλογές και γι' αυτό το λόγο Έχουμε ακούσει διάφορες ομιλίες με διάφορες αποχρώσεις έννοιες και θα συνεχιστεί αυτό. Θα ακούμε διάφορα ε, δεξιά και, αριστερά γιατί όλοι σκέφτονται τις εκλογές και θέλουν να υιοθετήσουν το σωστό σημείο. Θέλουν να βρεθούν στο σωστό σημείο. Εγώ όμως έχω ένα ερώτημα που έχει να κάνει με το κράτος δικαίου. Σε ό,τι με αφορά, γιατί έχω συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχω συμμετάσχει και στην ψηφοφορία για την έκθεση αυτό, να σας πω ότι όλοι στήριξαν τη ρουμανική ε, αντιπροσωπεία. Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι παιχνίδι. Στην Επιτροπή για τον Έλεγχο του Προϋπολογισμού γινόταν λόγος για το γεγονός ότι η Ρουμανία είναι ε, στις τρεις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά το σύστημα προστασίας ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα και την αυστηρότητα των ποινών και ότι θα μπορούσαν να διδαχθούν άλλα κράτη-μέλη από τα εξαιρετικά συστήματα προστασίας των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων που έχουν υιοθετηθεί στη Ρουμανία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ιδέα να υπάρξει ένας μηχανισμός σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ένας μηχανισμός συνεργασίας και επαλήθευσης και εξακρίβωσης και ελέγχου που θα ισχύσει σε όλα τα κρατημέλη με πολύ συγκεκριμένε υποχρεώσεις, κυρώσεις, δικαιώματα και ούτε καθεξής. Και όταν λοιπόν προτάθηκε αυτή η ιδέα και κατατέθηκε στο τραπέζι, εγώ ήμουν από τους πρώτους που τη στήριξαν. Όμως, δυστυχώς, με μετελικές πλεοτροπολογίες, η τελική τύχη του κειμένου αυτού ήταν η εξή. Αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την απάτη με ευρωπαϊκό κονδύλια και ότι είναι σοβαρό πρόβλημα αλλά τελικά προστίθενται και πολιτικά κριτήρια. Και εκεί κάπου χαθήκαμε, ε, χάλασε το πράγμα. Γιατί δεν είναι κακά τα πολιτικά κριτήρια αυτά κάθε αυτά αλλά τι θα πει αυτό ακριβώς. Μπορεί να κανείς να βάλει 5, 10 ή 100. Μα ζητούν βαθμολόγιο, scoreboard. Οποιουσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εάν η χ κυβέρνηση ή το ψ κράτο μέλος παραβαίνει το, το τάδε κριτήριο ή τον άλλο οποιοδήποτε κανόνα. Αυτό δεν επιδέχεται ανάλυση ή ερμηνεών. Δυστυχώς όμως αυτό δεν συνέβη τελικά, δεν πέρασε. Και η τελική δύναμη του, του κειμένου ελαττώθηκε. Τίθενται και νομικά θέματα κατά τη γνώμη μου και ισχυρά γιατί ο ορισμός είναι εξαιρετικά ευρύς και ασαφής και άρα δεν είναι σκόπιμος και κέριος. Αυτό καταρχάς και δεύτερον ποιος θα κρίνει. Εμείς προτείναμε και στηρίξαμε την ιδέα ενός πάνελ ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Και εδώ για άλλη μια φορά ε, βρήκαμε μπροστά μας ισχυρή αντίσταση στην ιδέα, αυτό, στην ιδέα αυτή και ε, μα ρωτούσαν σε ποιον θα παρουσιάσουν την έκθεση αυτή οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Αφού είναι ανεξάρτητοι μπορούν να διαπιστώσουν πράγματα και ε, μπορεί κανείς να πει ότι ναι ή όχι ο τάδε κανόνας ε, καταστρατηγήθηκε ή το τάδε μέρο του κοινοτικού κεκτημένου. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρουμε ποιο θα είναι ο τελικό κριτής, Ποιο θα αποφασίσει αν έχει υπάρξει παράβαση ή μη. Εγώ εκτιμώ και θεωρώ ότι καμία χώρα δεν μπορεί να κρίνεται με βάση τα πολιτικά κριτήρια. Α πάρουμε το παράδειγμα των κάτω χωρών. Εάν αύριο Κάποιο αποφασίσει ότι πρέπει να ισχύσουν αυτά τα κριτήρια π.χ. στις κάτω χώρες, διότι έχει υπάρξει ένα τεράστιο σκάνδαλο ε, ξεπλήματος χρήματος το μεγαλύτερο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο π.χ. Τι σχέση γι' αυτό με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι κάτι τελείως ξεχωριστό, τελείως διαφορετικό. Δηλαδή μια ε, καθαρή διαφοροποίηση χρειάζεται να γίνει. Αυτή είναι και η άποψη της Επιτροπής για τον έλεγχο του προπολογισμού γιατί εκεί έχουν συντάξει διάφορες εκθέσεις και έχουν συγκεκριμένη τεχνική αξιολόγηση και είναι υπέρ ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την πρόληψη της απάτης. Όταν όμως μπαίνει η πολιτική στη μέση, περιπλέκεται το πράγμα, τα πράγματα είναι πολύ πιο ασαφή, πολύ λιγότερο προβλέψιμα και πολύ περισσότερο πολιτικά. Σε ό,τι με αφορά θεωρώ ότι αυτό δεν είναι καλό. Αυτή η Επιτροπή έχει δώσει μεγάλο αγώνα υπέρ της ε, συνοχής. Κατά την άποψή σας, ποια είναι η σχέση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ξέρω ότι είστε ένθερμοι υποστηρικτής αυτής της έννοιας της συνοχής. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο και την πορεία σας. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής μας, επιτρέψτε μου να συνοψίσω κάποια από τα ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζι για την ανάπτυξη των περιφερειών, για τις περιφέρειες, γιατί όλοι λειτουργούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Όλοι οι συντονιστές και οι πολιτικές ομάδες αποφάσισαν να αποστείλουν μια ειδική επιστολή στον πρόεδρο Ταγιάννη, ο οποίος υποτίθεται ότι πρέπει να τη διαβιβάσει στην Ρουμανική Προεδρία και στην συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών Γενικών Υποθέσεων και εκεί επιμένουμε να έχουμε μια ευρύτερη προσέγγιση στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων γενικότερα. Γιατί ο περιορισμός σε συγκεκριμένα μπλοκ διαπραγμάτευσης ή σε συγκεκριμένα πεδία διαπραγμάτευσης μας δίνει πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας έτσι. Και οφείλω να πω ότι η δική μας Επιτροπή έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει τα καθήκοντά μας. Έχουμε τελειώσει από τη Βουλγαρική Προεδρία. Υποσχεθήκαμε να έχουμε την έκθεση για το Ιντερνετ τον Ιανουάριο και θα γίνει αυτό. Έχει ήδη γίνει και εγκρίθηκε και το CPR και κοινέ διατάξει, κοινό κανονισμό ε, θα είναι έτοιμο για το Φεβρουάριο, θα έχει εγκριθεί στην Ολομέλεια. Επομένω, εμεί ω Επιτροπή έχουμε δουλέψει πάρα πολύ εντατικά και έχουμε φέρει σε πέρα στα καθήκοντά μας ε, στο ισολόκληρο. Τέσσερις μεγάλοι φάκελοι έχουν προετοιμαστεί εδώ στην Επιτροπή μας. Μέρος του μπλοκ για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις διαπραγματεύσεις. Ζητούμε λοιπόν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να κάνει και αυτό ε, ε, το κομμάτι της δουλειάς που του αναλογεί. Εμείς δουλέψαμε εντατικά, είμαστε έτοιμοι να μπούμε στις διαπραγματεύσεις και επιμένουμε να μας δοθεί μια ευκαιρία να διαπραγματευτούμε. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε προφορικά. Σας δίνω το λόγο κυρία Υπουργέ και σας παρακαλώ να προσπαθήσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις των μελών. Ευχαριστώ. Πολύ. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ θερμά για τις ερωτήσεις σας για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Λαμβάνω το ισχυρό μήνυμα που εκπέμπει η Επιτροπή σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι πάρα πολλοί φάκελοι έχουν ήδη υιοθετηθεί και εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως εκπρόσωπος της Ρουμανικής Προεδρίας προσπαθώ να σας πω και μπορώ να σας πω ότι καταβάλουμε εμείς κάθε δυνατή προσπάθεια να προχωρήσουν οι φάκελοι και στο Συμβούλιο και να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και να μπούμε σε διαπραγματεύσεις. Ε, καταρχήν μπορώ να σας πω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με εσάς είναι τεράστια επιτυχία το γεγονός ότι εγκρίνατε την έκθεση για τον ε, κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις σήμερα το πρωί. σα συγχαίρω θερμά για αυτή την ψηφοφορία. Εκ μέρου της Προεδρίας ε, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορώ να σας πω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τους τριμερεί διαλόγους με βάση την εντολή που έλαβε το Συμβούλιο από τα κράτη-μέλη. Στόχος για τους τριλόγους, για τους τριμερείς διαλόγους δηλαδή, είναι να είναι έτοιμο το Συμβούλιο να διαπραγματευτεί και να ε, ε, συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εύθετο χρόνο. για να έχουμε μια ομαλή μετάβαση μεταξύ της υφιστάμενης γενιάς προγραμμάτων και της επόμενης γενιάς προγραμμάτων, γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι εγκαίρως. Το δίδαγμα που αντλήσαμε από την ε, τρέχουσα προγραμματική ε, περίοδο ήταν ακριβώς αυτό, ε, να καταπολεμήσουμε τις καθυστερήσεις και να κινηθούμε πιο γρήγορα. Καλωσορίζουμε λοιπόν την έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων με εσάς και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο τεχνικό. Ως εκ τούτου και επομένως, ως Προεδρία Ρουμανική δεχόμαστε την εντολή για το CPR, για το πρώτο και το πέμπτο μπλοκ και μπορούμε να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατό για τα θέματα αυτά. Ως οδικός χάρτης πορείας, να σας πω ότι μπορεί να ξεκινήσουμε και με το μπλοκ 2, είναι αυτό πιθανό, υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα, αν υπάρξουν και οι συνθήκες που θα μας το επιτρέψουν. Ελπίζουμε ότι θα λάβουμε την εντολή ε, στην Κορεπέρ της 30 Ιανουαρίου και επίσης για το ERDF και για το Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής μπορεί να ξεκινήσει και ο τριμερής διάλογος για τα θέματα αυτά. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την εντολή που θα λάβουμε. Εμείς ως Ρουμανική Προεδρία προσπαθούμε να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι κατανοούμε πολύ καλά και ε, τις ανάγκες και τα ωφέλη που θα έχουν οι δικαιούχοι και πόσο σημαντικό είναι για αυτούς να πετύχουμε αυτούς τους στόχους για να μπορέσουν να υπάρξουν επενδύσεις και για να δημιουργηθεί ευημερία για τον Ευρωπαίο πολίτη. Προσπαθούμε λοιπόν να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και να κάνουμε ό,τι περισσότερο και καλύτερο μπορούμε για να επιταχύνουμε το ρυθμό μας. Κυρία Γκρέλ, σας ευχαριστώ θερμά για το έργο σας και για τα καλά σας λόγια. Σας συγχαίρω και εσάς και τον κύριο Νόβακοφ. Για τη δουλειά που κάνατε για αυτό τον φάκελο. Συγχαίρω όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βοήθησαν. Αλλά και τους εμπειρογνώμονες. Γιατί ξέρουμε ότι δουλεύουμε με εμπειρογνώμονε. Όμω το πολιτικό μήνυμα είναι χειρό, είναι στεναρό και πρέπει να ακουστεί και σα συγχαίρω γι' αυτό. Τώρα, Όσον αφορά στα συγκεκριμένα επιμέρους ερωτήματα του κυρίου Νόβακοφ, να πω ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο στα πιο σημαντικά σημεία έτσι ώστε η προγραμματική περίοδος να μπορεί να ξεκινήσει το 2021 χωρίς καμία καθυστέρηση. όπως σας είπα, για τα μπλοκ 1, 5 και ίσως το 2 και για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Τώρα, από εκεί και πέρα. Για να δω τις σημειώσεις μου. Η κυρία Τόμασετς με ρώτησε διάφορα πράγματα. Να σας ευχαριστήσω θερμά κυρία Τόμασετς για τη δουλειά σας, για το έργο σας, για τα λόγια σας. Ως Συμβούλιο σας διαβεβαιώ ότι θα πράξουμε τα δέοντα, αυτά που μας αναλογούν, θα κάνουμε αυτό το καθήκον μας, αυτό που πρέπει, για να έχουμε αμερόληπτη προσέγγιση. Και πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να σας ευχαρώ εσάς, αλλά και τον συνάδελφο, Υπουργό Γκαμπριέλα. Θα είμαι στον Ντουμπρόβνικ ως φίλος της Συνοχής εκπροσωπώντας τη Ρουμανική Προεδρία. Κύριε Μίλτεμπεργκ, στρέφομαι σε εσά για να σας πω ότι βεβαίως τα συζητήσαμε αυτά και στο Βουκουρέστι. Ως προς το NEGO Box, το κοιτίο διαπραγμάτευσης για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι διατάξεις είναι αυτές που έχουν αναγνωριστεί και ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί από την προηγούμενη Προεδρία και την χάνουν ευρεία στήριξη από τα κράτη-μέλη. Άρα θα χρειαστεί πολιτική καθοδήγηση από τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων έτσι ώστε να μπορεί και το Συμβούλιο να καταλήξει στη δική του θέση. Η έκθεση του Συμβουλίου ευθυγραμμίζεται πλήρως με το ρόλο που έχει το Συμβούλιο βάσει των διατάξεων ε, που, της συνθήκης που ε, περιγράφουν το ρόλο του Συμβουλίου. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες έτσι διαμορφωμένες που να διαπροσωπεύουν και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των πολιτικών ηγετών. Το Κοινοβούλιο θα είναι στενά συνδεδεμένο στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα έχει την ευκαιρία πολλές φορές να εκφράσει την άποψή του, λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων σε αυτό το στάδιο. Το, το Συμβούλιο δεν είναι σε έτοιμο να διαπραγματευτεί με το Κοινοβούλιο για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι διαπραγματεύσεις αυτές πάντοτε γίνεται αντικείμενο συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών ηγετών και οι συνομοθέτες πάντοτε ήταν σε θέση και κατάφεραν να, να φτάσουν σε συμφωνία. Το φθενόπορο λοιπόν, φέτος του 2019, θα υπάρξει συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως γνωρίζετε. Ένα άλλο ερώτημα τώρα πώς σχεδιάζουμε τον τριμερή διάλογο για το Interreg και για τον κανονισμό για το Interreg και το CBM. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο έχει διαφορετική διαδικασία κάπως σε σχέση με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαφορετικές ομάδες στο Κοινοβούλιο συγγράφουν την εντολή αναλόγως, ενώ στο Συμβούλιο έχουμε ένα φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για τις διαπραγματεύσεις και για το Ίντερεκ και για το CBM. Είχαμε εστιάσει στα βασικά στοιχεία του πακέτου συνοχή που έχουν σχέση με το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν τι προετοιμασίε του για τα επόμενα προγράμματα. Επομένως, δεν ήταν δυνατό και εφικτό για το Συμβούλιο να έχει εντολή διαπραγμάτευση στις αρχές Ιανουαρίου για το Ίντερεγ και για αυτό το μηχανισμό του ECBM. Και άρα γι' αυτό η Ρουμανική Προεδρία δεν μπόρεσε να ξεκινήσει τριμερή διάλογο για τους φακέλους αυτούς. Οι μόνες εντολές που έχουμε είναι για αυτά τα μπλοκ που σας ανέφερα, το 1, το 5 και ίσως το 2. Και θα προσπαθήσουμε στο Συμβούλιο να κινηθούμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Για το μπλοκ 2, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Τι άλλα μπορώ να πω. για αυτά που είπαν ο κύριος Μίλτεμπερ και ο κύριος Νίκα για τη σχέση μεταξύ του κράτους δικαίου και της πολιτικής συνοχής. Εκ μέρους του Συμβουλίου θα συνεχίσουμε να ζητούμε την άποψη της νομικής υπηρεσίας όπως αυτό ζητείται από τα κράτη-μέλη και να την ακολουθούμε. Πολλοί γνωρίζετε ότι οι απόψεις αποκλίνουν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισχύει αυτό και συμβαίνει, άρα την απόφαση μπορούν να πάρουν μόνο οι ηγέτες, γιατί αποτελεί μέρος του Nego Box. Κύριε Μπούντα, απευθύνομαι σε εσά και θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Σε σχέση με την απλούστευση, Προφανώς, η πρόταση της Κομισιόν για την απλούστευση και την ευελιξία είναι εξαιρετικά ε, σημαντική. Όμως αυτή η διαδικασία είναι σε μια διαρκή εξέλιξη και για να αυξήσουμε το ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σκόπος της απλούστευσης είναι κυρίως να απλουστεύσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, έτσι. Και να λάβουμε υπόψη επίσης και την εθνική κλίμακα. Όλα εξαρτώνται από τη θέση των δικαιούχων. Συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία απλούστευσης, τηρώντας πλήρως τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Εδώ δεν εκπροσωπώ το Συμβούλιο. Να σας πω παρεθετικά ότι στη Ρουμανία ξεκινήσαμε τη διαδικασία το 2010 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και είναι κρίμα αυτή την παρένθεση δηλαδή τι κάνω μη εκπροσωπώντας το Συμβούλιο, μιλώντας προσωπικά και θα πρέπει να έχουμε μια συνολική θεώρηση κάθε εθνικής νομοθεσίας και να εξακριβώσουμε και να ελέγξουμε όλους τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να ε, βεβαιωθούμε και να μεριμνήσουμε έτσι, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές διατάξεις να τηρούνται στο σύνολό τους εις ολόκληρον. Διότι πρόκειται για ε, δημόσια έσοδα, για έσοδα του κρατικού κορβανά και θα πρέπει να δαπανώνται τα κονδύλια αυτά με ορθό τρόπο, με διαφανή τρόπο και γι' αυτό έχουμε αυτούς τους μηχανισμούς εξακρίβωσης, ελέγχου, audit. Και παρενθετικά να σας πω ότι στη Ρουμανία έχουμε ένα νόμο ο οποίος ισχύει και ο οποίος διέπει τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι έλεγχοι για να καταπολεμούμε την απάτη και αυτό είναι σημαντικό. Και έχουμε και τη δική μας ειδική διαδικασία για ό,τι έχει να κάνει με την ε, θέση της ελεγκτικής αρχής η οποία ε, ελέγχει μονίμως τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται οι δημόσιοι πόροι. Έρχομαι τώρα στο θέμα των προτεραιοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένη θέση έναντι ε, πλειάδας εθνικών διατάξεων όμως στηρίζουμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών ή των νομοθεσιών που έχουν να κάνουν με τις διοικητικές διαδικασίες. Σχετικά με το Interreg, έγιναν ήδη κάποιες επαφές στο Συμβούλιο, στα πλαίσια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, Οι συζητήσεις για τα θέματα σύνοχης δείχνουν ότι η αρχιτεκτονική την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αλλάξει. Και ότι η αντίληψη γύρω από τη δημιουργία ενός δικτύου είναι αυτή η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Σε συνεργασία με τους υπάρχοντες μηχανισμούς για τα διαμεθοριακά, ο κανονισμός αυτός, όπως είπατε, δεν συνδέεται με το CFP. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά θεσμικά θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα και αυτό θα απαιτήσει χρόνο. Αλλά νομίζουμε ότι επιμέρους θα βρούμε κάποιες λύσεις μέχρι το τέλος του μηνός Ιουνίου. Διακόπτει η κυρία Πλάμπ. Και την κυρία Ζωανά. Θα συμφωνήσουμε μαζί σας για την ανάγκη ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνέργεια ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνειδητοποιούμε την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να βελτιστοποιήσουμε τη συμπληρωματικότητα των πολιτικών και να αποκαταστήσουμε ένα ανεκτό επίπεδο χρηματοδότησης για την πολιτική συνοχής. Ένα άλλο ερώτημα σχετικά με τις τοπικές αρχές την έθεσε ο κύριος Μπούντα. Κατάλληλοι εταίροι είναι κρίσιμο για μας, είναι κρίσιμο για τις κυβερνήσεις, είναι κρίσιμο για το σύνολο της διαπραγμάτευσης και των διαβουλεύσεων. Mr. Για τον κύριο Νίκα. Nica. Da, Υπάρχει μια, ένας δεσμός ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την πολιτική συνοχής. Η αναχώρα συστάσεις το 2019 θα περιλαμβάνουν μέχρι το 2024 και ένα παράρτημα στα πλαίσια του οποίου οι επενδυτικές ανάγκες για κράτη-μέλη θα εγγράφονται αναλυτικά, έτσι ώστε το συγκεκριμένο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περίοδου να λαμβάνει υπόψη και τον προγραμματισμό των ταμείων και τις ενδιάμεσες αναθεωρήσεις. Υπάρχει επίσης και ένα νέο μέσο ενίσχυσης των ε, μεταρρυθμίσεων των διαφορετικών. Προβλέπονται ε, νέοι τρόποι χρηματοδότησης ε, των μεταρρυθμίσεων αυτών, χρηματοδοτήσεις συμπληρωματικές των υπολείπων ταμείων στην τομέα της διαφορετικής πολιτικής. Νομίζω ότι έχω απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες. Να σας ευχαριστήσω και για την υποστήριξή σας. Είμαι πεπισμένη ότι θα καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Ξέρω ότι και η δική σας εντολή ολοκληρώνεται ουσιαστικά στο τέλος Μαρτίου. Αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ε, για τον μήνα Μάρτιο. Για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική προς όφελος των πολιτών. Thank you, Ευχαριστώ την κυρία Πλούμπ και τις λεπτομερείς απαντήσεις. Ευχαριστώ και για την ενημέρωση για τα σχέδια του Συμβουλίου να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ε, και να μεταφέρετε το μήνυμα της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων προς το Συμβούλιο ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτες και οι τελικές ρυθμίσεις όπως είπατε για τις μελλοντικές νομοθετικές αποφάσεις γίνονται μέσα από κοινή απόφαση. Δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από το Συμβούλιο οι ρυθμίσεις αυτές. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σας εύχομαι κάθε καλό. Thank you, uh, dear colleagues. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Το επόμενο σημείο μας είναι η ανταλλαγή απόψεων με την uh, επίτροπο. Θα ελέγξουμε αν είναι εδώ θα ξεκινήσουμε αμέσως. Αν δεν είναι ακόμα εδώ θα, θα συνεχίσουμε σε 15 λεπτά. Okay, ladies and gentlemen, now we can continue with our meeting. Να συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι. Καθίστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το πρόγραμμα μας για τις ε, διαθεσμικέ ανταλλαγέ σήμερα το απόγευμα. Συνεχίζεται και τώρα έχουμε τη συζήτηση με την Επίτροπο Κρέτσου. Η επίτροπο λοιπόν ήρθε στις 31 Μαΐου στην Επιτροπή μας η τελευταία φορά. Έχει μεσολαβήσει λοιπόν μεγάλο διάστημα κατά το οποίο εργαστήκαμε ξεχωριστά. Και τώρα λοιπόν έχουμε πλέον αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε τις εξελίξει στην Επιτροπή Ρέτζη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής ε, εγκρίναμε την έκθεση μας από το Interreg στις 3 ε, Δεκεμβρίου στην Επιτροπή τον κανονισμό κοινών διατάξεων ε, σήμερα το πρωί. Και η Ολομέλεια ήδη έχει εγκρίνει το και Ελπίζουμε ότι και η σημερινή ψηφοφορία θα προγραμματιστεί για την Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. εγκρίναμε την, το μηχανισμό για τα διασυνοριακά εμπόδια και συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι το Φεβρουάριο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή την έκθεση για τα περιφερειακά ταμεία και τα ταμεία συνοχής. Η Επιτροπή έτσι λοιπόν εργάζεται σκληρά. Και θέλουμε να υποβάλουμε τις γνωμοτήσεις μας. Είμαστε έτοιμοι για τις θεσμικές ανταλλαγές. Σε κάποια από τα θέματα αυτά είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δε ανταλλαγή απόψεων με την Ρουμανική Προεδρία. Λίγο πριν από την άφηξή σας. Ελπίζω λοιπόν, Επίτροπε, ότι θα μας δώσετε μια πρώτη εκτίμηση για την έκτασή μα και για την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσο συνήθως ε, είμαι σίγουρη ότι θα είναι Πολύ ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, του βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και καταρχά θα ήθελα να σα ευχηθώ ότι καλύτερο για τη νέα χρονιά, η οποία είναι φυσικά ε, μεστή προκλήσεων. Σα εύχομαι κάθε ευτυχία και επιτυχία και σε εσά και στην οικογένειά σα. Δεν έχουμε βρεθεί εδώ και από πολύ καιρό, βέβαια, αλλά είχαμε και αυτή την ε, τριμηνία συνάντηση τον Οκτώβριο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την ε, έγκριση της έκθεσης CPR και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μεγάλο ορόσημο για τις διαπραγματεύσεις για το 2020. Είναι πραγματικά υψηλής ποιότητας και ε, την καταρτίζονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαστε ευγνώμονες που εργαστήκατε τόσο σκληρά. Δεδομένου δε το γεγονός ότι ήταν και χιλιάδες οι τροπολογίες που κατατέθηκαν Συγχαρητήρια. Και ευχαριστούμε. Καταρχάς πρώτα προς την Κωνσταντσα και τον Αντρέη, αλλά και σε όλους σας και στους υπαλλήλους και βοηθούς. Είστε άξιοι επένων. Καλώς ορίσω και την υποστηρίξή σας για τις δεύτερες γραμμές της μεταρρύθμισής μας. Εξυγχρονισμό, εμβελεξία και απλούστευση. Καλώς ορίζω και την υποστήριξη για τα νέα επιτεύγματα της πολιτικής, ε, τα ανανεωμένα προγράμματα αλληλικής σχέσης, ε, η ενισχυμένη προσέγγιση περιφερειακής διάστασης και η διαχείριση και τα συστήματα ελέγχου. Κατα... Χαίρομαι για την υποστήριξή σας για την πολιτική για τον προπολογισμό και χαίρομαι που έχετε ακόμα εμπιστοσύνη για την πολιτική μας που χρειάζεται χρειάζεται για τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Η οικονομική και περιφερειακή πολιτική θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής, του ευρωπαϊκού έργου. Η έκθεση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, όπως ε, και η έκθεση Interreg που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια. Να συγχαρώ τον εισηγητή και τους κοιότητες εισηγητές. Είναι πολύ καλή η έκθεση αυτή. Και τώρα είναι η στιγμή να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Αν θέλουμε να αποφύγουμε τις ε, καθυστερήσει σε ό,τι αφορά την περίοδο μετά το 2020, θα πρέπει να εγκρίνουμε τον κανονισμό φέτος. Το είπαμε ευθύ εξ αρχή ότι θα πρέπει να γίνει αυτό πριν από τις ευρωεκλογέ. Ξεκινάνε λοιπόν τώρα οι τριμερεί διάλογοι και φαίνεται ότι υπάρχει πλέον αυτή τη δυνατότητα. Είναι πραγματική αυτή η δυνατότητα. αν δεν εγκρίνουμε τον προπολογισμό και τον κανονισμό μέχρι το τέλη του έτους, ε, ρισκάρουμε να χάσουμε χρόνο και δεν θα προλάβουμε να καταστούν λειτουργικά τα προγράμματα από 1η Ιανουαρίου 2020. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε ακριβώς αυτό το στοιχείο, να αντιδραματίσουμε το ρόλο μας και να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Ευρωπαϊκός Προλογισμός για τους πολίτες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τους τριμερείς διαλόγους και τις συζητήσεις έχετε δώσει ένα νέο έναυσμα με την έκθεση αυτή, μπορούμε θεωρώ να ξεκινήσουμε άμεσα. Σας ζητώ λοιπόν και από εσά και από τη Ρουμανική Προεδρία να μην κόψετε ταχύτητα και να έχετε διάθεση στους τριμερείς διαλόγους. Να διατηρήσουμε λοιπόν αυτή την ορμή, αλλά και την ποιότητα των προτάσεων για μια αποτελεσματική και σύγχρονη πολιτική συνοχή. Να σα υπενθυμίσω κάποια βασικά στοιχεία τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να διατηρηθούν. Και ασφαλώ τη δική σα υποστήριξη να εξασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αποδυναμωθούν τελικά στι διαπραγματεύσει. Το πρώτο λοιπόν βασικό στοιχείο είναι η Συμφωνία Εταιρική Σχέσεω για όλα τα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιε απόψει για να προσθεθούν κάποια κράτη-μέλη και όχι κάποια άλλα η έκτασή σας σωστά επισημαίνει τη στρατηγική βάση της πολιτικής μας ε, για το θέμα του συντονισμού και για τις συνέργειες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Πιστεύω ακράταντα ότι όλες ε, οι χώρες θα πρέπει να έχουν στρατηγική προσέγγιση και εταιρική σχέση, ακόμα και χώρες με μικρή, μικρά ποσά, ακόμα και με χώρες για με κυβερνητικά προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ισχυρή στρατηγική βάση για τα κρατημέλη που παρουσιάζουν τους στόχους και τα αποτελέσματα που αναμένονται. Τα θέματα αυτά, ξέρετε, δεν είναι τεχνικά. Θεωρώ ότι είναι θεμελιώδη και είναι θεμελιώδης επιλογές σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές πολιτικές. Και έτσι, λοιπόν, δεν δημιουργείται επίσης επιπλέον γραφειοδοτικό άχθος. Μία σημαντική επιλογή είναι ο συντονισμός των ταμείων. Πιστεύω απόλυτα ότι σε μια πλήρη τέτοια πρόταση εταιρική σχέση προτείνουμε 7 ταμεία στο CPR για να υπάρχει καλύτερο στρατηγικό επίπεδο και εφαρμογή σε ό,τι αφορά τα ταμεία και σε ό,τι αφορά και τις 27 χώρες. Κατά την απόψή μας δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ε, διπλά μέτρα και σταθμά, διαφορετικούς κανόνες για διαφορετικά κράτη-μέλη ούτε διαφορετικούς κανόνες για διαφορετικά ταμεία. Και όπως είπα στην αρχή, ελπίζω πραγματικά να έχω την υποστήριξή σας στο θέμα αυτό. Δεύτερο σημείο κλειδί, το θέμα του προγραμματισμού 5 συν 2. Σας ενθαρρύνω να δείξετε ανεκριτό πνεύμα, γιατί εδώ θεωρώ ότι θα έχει νόημα αυτή η ενδιάμεση θεωρή, αν σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοδότηση εξ αρχής. Αυτό μειώνει την ευελιξία και η εμπειρία δείχνει ότι αυτό είναι κακό για να ανταποκριθούμε στις ε, προκλήσεις. Για παράδειγμα, την προηγούμενη πραγματική περίοδο δεν περιμέναμε την μεταναστευτική κρίση και κληθήκαμε να αλλάξουμε πάρα πολλά προγράμματα τελικά εκ των υστέρων και σε κάποια κράτη-μέλη. Έγινε μεταφορά των πόρων διότι δεν είχαν επαρκή προγράμματα σε κάποιε τομεί. θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία στην ενδιάμεση αθαερόριση. Ανάλογα με τι ε, ανάγκες των πολιτών. Αν διαγράψουμε το 5 συν 2, θεωρώ ότι θα κάνουμε ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά την ευελιξία και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ο προγραμματισμό 5 συν 2 είναι κακός για τα μακροπρόθεσμα έργα. Δεν είμαι πεπισμένη τα μακροπρόθεσμα έργα θα παραμείνουν στο επίκεντρο της πολιτικής ε, συνοχής, θα είναι τμήμα της ενδιάμεσης αναθεώρησης, θα μπορούν να επιλεχθούν ε, νωρίτερα στη διαδικασία και ακόμα και για έργα που θα εφαρμοστούν μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση θα έχουν τέσσερα έτη. Ουσιαστικά είναι 5 συν 4, δεν είναι 5 συν 2 τα χρόνια. Γιατί οι δαπάνε μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος του 2029. Άρα από το 5 συν 2 θεωρώ ότι εγγυάται μεγαλύτερη ευελιξία για τις δαπάνες και δεν αποτρέπει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Το τρίτο θέμα κλειδί, θεματική επικέντρωση. Ο συνάδελφος ο κ. Κοτσολίνο εργάζεται σκληρά για το θέμα των Ταμείων Συνοχής στη σχετική γνωμοδότηση και προσβλέπω στο τελικό αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ θα ήθελα να πω ότι οι προτάσεις μας για την θεματική επικέντρωση είναι πολύ φιλόδοξες. Οι στόχοι μας ε, είναι πολύ φιλόδοξοι και από πλευρά του υπολογισμού θα πρέπει να επιδείξουμε υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας για να κινηθούμε προς μια ευφυή ε, Ευρώπη χαμηλού άνθρακα, ψηφιακή και είμαι πεπισμένη ότι αυτέ είναι οι δικασίες απαραίτητες. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μεγάλη ευελιξία στην θεματική επικέντρωση να ληφθούν ελευθερά τις περιφερειακές συνθήκες υπόψη. Επίσης, η ευελεξία θα πρέπει να καλύψει διάφορες διαφορετικές προκλήσεις. Για παράδειγμα, στις περιοχές εντατικής χρήσης άνθρακα. Θεωρώ ότι το Ταμείο για την Ενεργειακή Μετάβαση θα διευκόλυνε τη μετάβαση και κυρίως ό,τι αφορά τις περιοχές άνθρακα εδώ βλέπουμε όμως κάτι διαφορετικό, ότι δεν λείπουν οι πόροι, λείπει η διοικητική διαχείριση. Αυτό αποτρέπει την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και των έργων. Και να πω επίσης ότι η πολιτική συνοχή είναι κάτι ήδη γνωστό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα νέο τομείο θα δημιουργήσει προβλήματα ουσιαστικά και σύγχυση στους δικαιούχους. το σημείο κλειδί. Το θέμα τη απλούστευση, εγκάρσιο θέμα. Σα ευχαριστώ εδώ για την υποστήριξή σα και ξέρετε καλά ότι ήμουν υπέρ τη ριζική ε, απλούστευση. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην κοινή αυτή προσπάθεια για την απλούστευση, γιατί πολλέ από τι προτάσει απλοποίηση βασίζονται σε ιδέε και προτάσει από όλα τα μέλη της ε, οικογένειας συνοχή. Ε. Απλοποίησαμε τα προγράμματα, την κατάρτιση των πραγμάτων, τη διαδικασία ελέγχου, Υπάρχει μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανόνων σε όλα τα ταμεία. Έχουμε ενιαίους κανόνες για τις επιδοτήσεις και τα οικονομικά μέσα και έχουμε ένα εγχειρίδιο 80 μέτρων μέσων ε, απλοποίησης. Σας ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξή σας, για τις προτάσεις αυτές. Ξέρετε καλά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ της απλούστευσης αυτής. Φυσικά η απλούστευση δεν είναι αυτός σκοπός η ευελιξία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο τελικός στόχος είναι η συνοχή. Η ευελιξία και η απλοποίηση είναι ένα μέσο μόνο. Απότερο στόχο θα πρέπει να είναι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας. Αυτή η αποτελεσματικότητα λοιπόν υποστηρίζεται από σχέσεις, από την απλούστευση, από την θεματική επικέντρωση. Αυτή είναι η πυλώνα μια αποτελεσματικής πολιτικής, θεωρούμε. Θα πρέπει να εμπεριθούν λοιπόν αυτοί οι πυλώνες αν θέλουμε να, να υποστηρίξουμε το κτίσμα. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την υποστήριξή σας και ζητώ να συνεχιστεί αυτή και στις υπόλοιπε πολιτικές. Στου τρει μερίδε διαλόγου για να ολοκληρωθούν γρήγορα και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε τι εργασίε μα τις ε, κοινέ όσο πιο γρήγορα γίνεται. για τις διαπραγματεύσεις τον Απρίλιο. Τα πιο σημαντικά στοιχεία σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα μετά το 2020 είναι οι διαπραγματευτικέ εντολέ των δύο συνομοθετών και έχω υπόψη μου το θέμα του προγραμματισμού και τη διαχείριση του ελέγχου. Ένα τρίτο αυτό αποτελεί του κανονισμού. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνο να συνεχίσουμε στην παρούσα φάση. Ξέρουμε ότι δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα μέχρι ότου συμφωνηθούν τα πάντα, προφανώ. Αυτό θα δώσει όμως μια στεναρή βάση για το επόμενο κοινοβούλιο επί τη οποία θα μπορέσουν να εργαστούν και θα δώσουν μεγαλύτερη σαφήνεια και στις αρχές διαχείρισης στην κάθε χώρα. Ήδη λοιπόν θέτεται τον σχετικό ρυθμό και σε ό,τι αφορά τις προτάσεις CPR και τους υπόλοιπους κανονισμούς. Ασφαλώς θα πρέπει να ασκήσουμε επίσης στο Συμβούλιο για να βιαστούμε μέχρι τον Απρίλιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία και προσβλέπω στη συνεργασία. Σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας. Uh, ευχαριστώ πρώτα τις ερωτήσεις και για τον τριμερή διάλογο. Είχαμε συνάντηση, ξέρετε, με την εκπρόσωπο της Ρουμανικής Προεδρίας και συζητήσαμε το θέμα των τριμερών διαλόγων και θα το συζητήσουμε και με εσά. Η κυρία Κρέλ πρώτα, παρακαλώ. Νόμιζα ότι θα ξεκινήσουμε με τους συντονιστές, λέει η κυρία Κρέλ. Αλλά όπως θέλετε. Βεβαίως και να ξεκινήσω πρώτη-πρώτη. Κυρία Πίτροπε, Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαστε εδώ πάλι στην Επιτροπή μας. Και είναι και ευτυχή η σημερινή ημέρα, γιατί σήμερα ολοκληρώσαμε τη δύσκολη ψηφοφορία για το CPR. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί επίτευγμα για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι όλους όσοι συνέβαλαν στην ε, επίτευξη αυτού του καλού αποτελέσματος. Πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή στεναρή βάση για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Τα θέματα τα οποία αναφέρατε. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο είναι πάντα από, στην πλευρά της ε, Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις ε, συμφωνίες Εταιρική Σχέση και την αρχή τη εταιρική σχέση, όπω την αναφέρατε, σχετίζεται στενά. Τα υποστηρίζουμε όλα αυτά και θέλουμε ασφαλώ να τα ενισχύσουμε. Από δική μου πλευρά, θα αποτελέσει αυτό σημαντικό στοιχείο και στους τριμερείς διαλόγους για το Κοινοβούλιο. Προς αυτή την πλευρά θέλουμε να διαπραγματευτούμε. Και εννοείται ότι υποστηρίζουμε και την Επιτροπή στην προσφορά που κάνει για απλοποίηση της πολιτικής ως ε, συνηγήτρια από κοινού και με τους κοιόδες εισηγητές θα ήθελα να πω ότι μου επισημάνθηκε ότι δεν έπρεπε να γίνουν τροπολογίες ε, οι οποίες τελικά θα είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή επιπλέον ε, προδιαγραφών. Ελπίζω να το πετύχαμε αυτό. Από την άλλη, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φυσικά θα ήθελα να έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες ε, σε ό,τι αφορά το θέμα της εξέλιξης του θέματος του φύλου στα κράτη-μέλη. Και εν μέρη είχαμε κάποιες σχετικές τροπολογίες και ω εισηγητέ μιλήσαμε για το θέμα αυτό, γιατί ξέρουμε ότι θέλουμε να γίνει συλλογή των δεδομένων αυτών και ότι είναι μεγάλο όμω τελικά το γραφειοκρατικό άκθο που συνεπάγεται αυτό το μέτρο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να επιλέξουμε την οδό τη απλούστευση σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή. Έχουμε επίση ε, ψηφίσαμε μάλλον με μεγάλη πλειοψηφία σε ό,τι αφορά τις ε, μεταφορές μεταξύ διαφορών ταμείων και διαφορετικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε αυτό να δημορφωθεί με τόσο γενναιόδωρο τρόπο όσο πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί, γιατί θεωρούμε ότι μετά από τις ε, επίπονες ε, ε, περικοπέ που αναγκάστηκε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τον τομέα τη πολιτική συνοχή, δεν μπορούμε να παριστάνουμε Απλά λες και έχουμε αυτόν χρήμα για να μεταφέρουμε και σε άλλες, σε, σε άλλους τομείς, σε άλλα προγράμματα από το Connecting Europe Facility. Θεωρώ ότι ο συμβασμός που πετύχαμε είναι καλός σε ό,τι αφορά τις μεταφορές αυτές και για τις ε, συνεισφορές σε άλλα προγράμματα. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποστηρίξει και στην διαπραγματεύση με το Συμβούλιο. Γιατί αυτό που απασχολεί την Επιτροπή μας είναι να έχουμε με ευελιξία αφενός, αλλά από την άλλη να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς είμαστε οι αρμόδιοι για την προάσπιση στη τελική ανάλυση της πολιτικής συνοχής. σε ό,τι αφορά το ERDF και το Ταμείο συνοχή και στο σχετικό κανονισμό δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει τι εργασίες μα, άρα δεν μπορώ να αποφανθώ επ' αυτού. Ελπίζω μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου να μπορέσουμε να ψηφίσουμε με το καλό στην Επιτροπή μας, να συγκεντρώσουμε και να καταρτήσουμε συμβαστικές προτάσεις. Δυστυχώ, οι εργασίε για το Interreg που ολοκληρώθηκαν στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα προφανώ δεν μπορεί να οργανώσει την σχετική εντολή το Συμβούλιο για να ξεκινήσουμε τις τριμερεί διαλόγους και είναι κρίμα γιατί αυτή η συνοριακή συνεργασία είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερω τους Ευρωπαίους πολίτες και είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει πραγματική ευρωπαϊκή υπεραξία στα σύνορα. Σε ό,τι αφορά την διασυνοριακή λοιπόν, συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι γίνεται απτή, πραγματικά απτή και θα Ήθελα πολύ να μπορούσα να ξεκινήσω την διαπραγματεύσει. Για το CPR αυτό που μπορώ να πω είναι το εξή. Θεωρώ ότι θα λάβουμε το Φεβρουάριο στην Ολομέλεια την εντολή. Ελπίζω χωρί μεγάλε αλλαγέ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε αυτό. Και ελπίζω παρά αυτά να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με τον τριμερή διάλογο. Η Προεδρία ανέφερε και είπε ότι έχει ολοκληρώσει δύο ενότητες σε ό,τι αφορά την εντολή και ενδεχομένω ε, να μπορέσει να υποβάλει και άλλα τμήματα σε ό,τι αφορά την εντολή. Αν καταφέρουμε λοιπόν το θέμα του προγραμματισμού και της διαχείρισης να το διαπραγματευτούμε από κοινού, θεωρώ ότι αυτό ήδη θα αποτελέσει ένα σημαντικό μήνυμα προς τις ε, περιφέρειες και προφανώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ελεύθερο στη λήψη αποφάσεων του, αλλά νομίζω ότι όπως και να το κάνουμε ένα νέο ε, νέο εκλεχθέν κοινοβούλιο του, οποίου το σύνθεση φυσικά δεν γνωρίζω ακόμα, θα εκτιμήσει τη δουλειά που θα του υποβάλουμε, γιατί νομίζω ότι και το νέο κοινοβούλιο θα συνειδητοποιεί ότι από 1η Ιανουαρίου του 2020-2021 θα πρέπει να έχουμε μια νέα πολιτική η οποία να είναι λειτουργική και άρα αξίζει τον κόπο όλοι να καταβάλουμε την προσπάθεια για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε σωστή υποστήριξη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Very much. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τώρα με τους συντονιστέ. Κύριε Τόμασιτ, έχετε το λόγο. Η κυρία Τόμασιτ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, καλωσορίσατε στην ε, συνεδρίασή μας. Έχω ένα ερώτημα το οποίο με απασχολεί από τότε που πρώτο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εύκολο να το θέτει κανείς, δύσκολο να το απαντά. Με βάση την εμπειρία σας, πώς μπορεί να βοηθήσει η Επιτροπή και να ενθαρρύνει τα κρατημέλη και μάλλον στα τα λιγότερο ανεπτυγμένα κρατημέλη, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στις σημαντικές νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς η πράξη μας διδάσκει ότι η καλή γνώση των κανόνων ε, δίνει τη δυνατότητα σε ορισμένα κράτη-μέλη να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενώ όσοι είναι λιγότερο ενημερωμένοι και λιγότερο ενεργοί και δραστηροί, δεν έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ίσως δεν είναι καθήκον αυτό της Επιτροπής θα μας πείτε, αλλά εγώ νομίζω ότι η Επιτροπή είναι τόσο καλή όσο είναι το πιο αδύναμο κράτος μέλος. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλωσορίσατε κυρία Επίτροπε, λέει ο κύριος Μίλτεμπεργκ. Συζητήσαμε το CPR, το κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις και ένα από τα βασικά θέματα είναι η δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων από ε, τα διαρθρωτικά ταμεία στα ταμεία που γίνονται αντικείμενο άμεσης διαχείρισης και διοίκησης. Και προτείναμε κάτι πολύ πιο αποδυναμωμένο. Μας εξηγείτε γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό να έχουμε τη δική σας συνεισφορά το συζητήσαμε και στην Ολομέλεια και πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα να υποβάλουμε τροπολογίες. Αυτό είναι καταρχάς το πρώτο μου ερώτημα. Από εκεί και πέρα πήραμε όλες τις πληροφορίες και ξέρουμε τι γίνεται με τις αποδεσμεύσεις. Γιατί η Ρουμανία υπήρχε σοβαρό κινδύνος αποδέσμευσης να χαθούν τα κονδύλια. Ε, και το είπατε ξεκάθαρα για τη Ρουμανία και είδα στη σελίδα σας στο facebook ότι οι ρουμανικές αρχές πρότειναν τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς έργα ύψους 629 εκατομμυρίων ευρώ. Ζήτω τα μέσα κοινωνική δικτύωσης, γιατί αλλιώς δεν θα τα είχαμε μάθει αυτά. Δεν είναι αυτό προβληματικό και από την πλευρά της προστατικότητας. Εάν τα κράτη-μέλη ουσιαστικά παρουσιάζουν project και προγράμματα τόσο αργά στο τέλος της χρονιάς, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και αμφιβολίες. Και από πλευράς ελεκτικού συνεδρίου, για το θέμα της προσθετικότητας επίσης. Ένα από τα έργα τα οποία λήφθη υπόψη ήταν η η απόκτηση 700 ασθενοφόρων. Πολύ σημαντικό αυτό για το ε, ρουμανικό ΕΣΥ, ε, για τον ε, τομέα της υγείας στη Ρουμανία, νέα ασθενοφόρα για να μεταφερθούν οι ασθενείς και όσοι χρήζουν νοσοκομιακής παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση όμως, σύμφωνα με τα δικά μου στοιχεία, θα αγοράζονταν χρησιμοποιώντας εθνικά ε, ρουμανικά κονδύλια. Άρα τίθεται το ερώτημα της προσθετικότητας Και το τελευταίο μου ερώτημα, σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο πάντοτε, δημοσιεύσαν μια έκθεση για την καταπολέμηση της απάτης και είδα ότι οι ανακτήσεις μετά από την εφαρμογή όλων των συστάσεων είναι πολύ χαμηλότερες στη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο από ό,τι στις άλλες γενικές διευθύνσεις. Στη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση ε, επανακτάται το 32%, στη Γενική Διεύθυνση για το Γεωργία 30 της εκατό, ενώ στη Γενική Διεύθυνση Ρέτζι ανακτούν μόνο το 10 της εκατό ε, αφού έχει διαπιστωθεί η διασπάθηση των κονδυλίων. Ίσως πρέπει να επιταχύνετε τις δράσεις σας για να ανακτάτε όσο δυνατόν περισσότερο και καλύτερα τα κονδύλια που διασπαθίζονται. Ο κύριος Παπαδημούλης παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, <clears throat> σας καλωσορίζω Επίτροπα Κρέτσου για μια ακόμη φορά στην Επιτροπή μας. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Ε, θα ήθελα να θέσω ορισμένα θέματα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι επόμενοι μήνες και ή δυνατόν πριν από τις ευρωεκλογέ έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και είναι μια ευκαιρία η Κομισιόν και η Ρουμανική Προεδρία να ανεβάσουν ταχύτητες γιατί αν αναβληθεί η συμφωνία σε αυτό το θέμα θα χάσουμε όχι μόνο χρόνο αλλά θα χάσουμε και χρήματα γιατί θα καθυστερήσει η προετοιμασία των σχετικών προγραμμάτων. Και αυτό θα έχει κόστος και οικονομικό και κοινωνικό σε μια περίοδο που η Ευρωζώνη κατεβάζει τους προβλεπόμενους ρυθμούς ανάπτυξης. Επομένως η ερώτησή μου η πρώτη είναι τι εκτιμάτε ότι θα γίνει. Θα παραπευθεί το θέμα στις καλένδες, θα έχουμε τον κίνδυνο μιας αναβολής, θα φτάσουμε στο 2020 χωρίς να έχουμε τις συμφωνίες για να αρχίσουν να, να προχωρούν τα προγράμματα. Το δεύτερο θέμα είναι το Interreg. Θα προλάβουμε αυτό το θετικό που ψηφίσαμε, το ανέφερε και η κυρία Κρέλ, στην ε, Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου να προχωρήσει, να ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος για να αρχίσουν να εφαρμόζονται αυτά τα προγράμματα. Σε δύο μέρες η χώρα μου η Ελλάδα επικυρώνει μια ιστορική συμφωνία με την πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας η οποία λύνει με θετικό τρόπο που τον χαιρετίζει και το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό και η Κομισιόν και το Συμβούλιο μια μακρά διαμάχη περίπου τριών δεκαετιών. Δεν μας αρκούν τα χειροκροτήματα της διεθνούς κοινότητας. Αν είχαμε και τα κονδύλια του Ίντερεγ για προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας θα ήταν πολύ καλύτερα για τους πολίτες και των δύο χωρών να δουν τις ορατές βελτιώσεις στη ζωή τους. Το τρίτο θέμα αφορά την απλούστευση. Ναι, συμφωνώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει βοηθήσει πολύ μαζί και με εσά στο να γίνουν βήματα απλούστευσης. Αλλά θα ήθελα λίγο να προσέξουμε και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για παράδειγμα, στην πρόταση της Κομισιόν για τη νέα πολιτική συνοχής στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχουν ληφθεί και σωστά και άλλα κριτήρια εκτός από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν για την κατανομή των κονδυλίων, όπως είναι κοινωνικά κριτήρια που έχουν σχέση με το ύψος της ανεργίας. Μπορείτε να μου πείτε γιατί για το CPR λαμβάνεται ως μόνο κριτήριο το ΑΕΠ και όχι και άλλα κοινωνικά ε, κριτήρια. Και επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά δύο πράγματα με λίγα λόγια. Το πρώτο, Έχω μια ανησυχία γιατί η ενσωμάτωση του Ταμείου Μετανάστευσης στο CPR δεν παίρνει υπόψη της το εξής γεγονός ότι οι προσφυγικές ροές βαρύνουν κυρίως τις χώρες υποδοχής γιατί έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν δίνει ευρωπαϊκές λύσεις στο προσφυγικό. Επομένως υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί από την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέμβει συνολικά, να επιβαρυνθούν πρόσθετα οι χώρες υποδοχής, όπως η χώρα μου η Ελλάδα. Και το δεύτερο, υποστηρίζω με έμφαση την διακριτή μεταχείριση των νησιών, γιατί τα νησιά και όσες χώρες έχουν έντονη νησιωτικότητα όπως η Ελλάδα, αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα προσβασιμότητας για τους πολίτες και τα αγαθά. Τέλος, η πολιτική μου ομάδα σκοπεύει με τροπολογίες, παρότι έγινε καλή δουλειά στο CPR, να επαναφέρει το θέμα της δημοσιονομικής αιρεσιμότητας, γιατί θεωρούμε λάθος να τιμωρούνται περιφέρειες επειδή ενδεχομένως οι κυβερνήσεις τους δεν κάνουν ορθή δημοσιονομική διαχείριση. Και τα λέω με την άνεση ότι η χώρα μου η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ενδεχομένως πιο νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά και από τη Γερμανία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπρέσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω, Επίτροπε. Δύο σημεία να θέσω. Το ένα το έθεσαν αρκετοί συνάδελφοι. πέρα από την πρόοδο στην οποία μπορεί να καταλήξει ο τριγωνικός διάλογος, δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε συνολικά αν δεν υπάρξει ποσοτική συμφωνία θέλετε και αυτό ισχύει για όλους τους κανονισμούς ουσιαστικά τους οποίους ε, συζητάμε σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε σε όλα τα πεδία, στο τέλος τίποτα δεν θα συμφωνήσουμε αν δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για τους αριθμούς τα πάντα. Πάνω σε αυτό το κοινοβούλιο ε, επιμένει. Επιμένει γιατί είναι η μοναδική δυνατότητα την οποία έχει το κοινοβούλιο να ασκήσει τις εξουσίες του. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι πρέπει να κάνετε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να προσπαθήσετε αν όχι να καταλήξουμε σε μια πλήρη συμφωνία πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου αλλά τουλάχιστον να μπορέσετε να κάνετε κάποια σημαντικά βήματα για μια συμφωνία που θα ονόμαζα συμφωνία πλαίσιο η οποία θα επιτρέπει να διαγράφονται κατά κάποιο τρόπο οι βασικές γραμμές και θα επανέλθουμε τον Οκτώβριο, γιατί βέβαια τον Οκτώβριο θα έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο και μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα είναι υποδιαμόρφωση, οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσει όλους τους κανονισμούς. Είναι σημαντικό δηλαδή τα βήματα προόδου ανεξαρτήτως της κατάληξης σε αυτή τη φάση να γίνουν αυτή την περίοδο. Τώρα μια δεύτερη ερώτηση πολύ πιο απλή από την πρώτη. Όλοι εμείς που προερχόμεθα από αγροτικές περιοχές, από περιφέρειες, από ορεινές, νησιωτικές κτλ. που αποτελούν ουσιαστικά το 80% του εδάφους της Ένωσης και το 40 50% ε, του πληθυσμού. Θα θέλαμε ε, να κλείσει και η δική σας περίοδος, θα θέλαμε να συνεχίσετε, αλλά τουλάχιστον θα θέλαμε να μας πείτε τι έχετε κάνει ε, ειδικά για τις ορεινές και απόμακρες περιοχές. Ιδιαίτερα γιατί μέσα από τον καινούριο κανονισμό, ο οποίος τίνει σε μια κάποια συγκέντρωση θα έλεγα και σε ευρωπαϊκού τύπου προσανατολισμούς ε, της χρήσης ε, των πιστώσεων αυτών καλό θα είναι να υπάρξει ε, ένας μεγαλύτερος αριθμός στόχων επιμέρους. Ας πούμε, η ψηφιακή ατζέντα. Η ψηφιακή ατζέντα δεν είναι το ίδιο πράγμα για μια αστική περιοχή και για τις ε, περιοχές της υπαίθρου. Ναι μεν ο στόχος είναι ένας, ναι μεν ο στόχος είναι ενιαίος, αλλά φυσικά η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου θα πρέπει να γίνει με διαφορετικούς τρόπους στις αστικές περιοχές και διαφορετικούς στις ε, περιοχές τις ορεινές, τις απόμακρες κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσετε να βοηθήσετε τις περιφέρειες ε, να πετύχουν τους στόχους στον τομέα της ψηφιακής ατζέντα. Περιμένουμε λοιπόν από πλευρά σας ε, κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας περίοδου και κατά τη διάρκεια και της ρωμανικής Προεδρίας να ξεκινήσετε μία προσπάθεια η οποία θα βοηθήσει να πετύχει τους στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο θεματολογικής συγκέντρωσης για όλα τα επιμέρους εδάφη της Ένωσης και όχι μόνο για συγκεκριμένα. Γιατί ακριβώς το πρόβλημα είναι ότι στις περιφέρειες οι οποίες έχουν αργούς ρυθμούς ανάπτυξη δεν καταφέρνουμε να προχωρήσουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς μένει όλο και πιο πίσω. Λοιπόν, θα ήθελα να μάθω σε ποιο βαθμό λαμβάνεται υπόψη τα ψηφίσματά μας μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νοβακόφ έχει το λόγο. Ως ε, εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συντονιστής μάλλον, ε, να σας ευχαριστήσω, όπως επίσης και σαν συνεισηγητής για το CPR. Σήμερα κλείσαμε όπως γνωρίζετε το πρώτο βήμα της διαδικασίας, καταλήξαμε σε μία πλειοψηφία με ισχυρή θα έλεγα στήριξη και ελπίζουμε να πάρουμε τη συγκεκριμένη εντολή και να ξεκινήσετε διαπραγματεύσεις άμεσα. Πριν από εσά, ήδη η αρμόδια υπουργός της Προεδρίας είπε ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες και θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι εμένετε και εσείς στην αρχική σας θέση. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν ποιες είναι οι βασικές αλλαγές τις οποίες προτείνετε θα έλεγα και αν λαμβάνετε υπόψη αυτά τα οποία λέμε εμείς για το CPR. Οι αποφάσεις τις οποίες πήραμε δεν ήταν εύκολες και δεν ήταν εύκολο να βρούμε τη σωστή διατύπωση για να υπάρξει απαιτούμενη στήριξη. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας για τις θέσεις αυτές. Είναι προφανές ότι έχουμε και άλλα θέματα τα οποία έχουν σημασία στο εσωτερικό της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μην επαναλάβω αυτά τα οποία είπε η κυρία Κρέλη, συνεισηγήτρια. Πάντως, για θέματα ποσοστού ε, συγχρηματοδότησης, για μεταφορές. Ε, ε, νομίζω μπορούμε να βρούμε κάποιο κοινό τόπο και να περάσουμε στην επόμενη περίοδο. Και εδώ σημασία έχει το χρονοδιάγραμμα, πότε μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ την Επίτροπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες τις οποίες έχετε κάνει μέχρι τώρα για τη στήριξη της πολιτικής συνοχής. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να περιοριστούμε στο να δώσουμε στα κράτη-μέλη κάποια έγγραφα τα οποία απλά θα περιλαμβάνουν, αν θέλετε, τον ορίζοντα τον οποίο θα έχουμε μπροστά μας για την πολιτική συνοχή. Θα ήθελα κάτι το πιο συγκεκριμένο να σας πω για τη δική μου χώρα. Πρόσφατα με το διάταγμα 114 οι αρμοδιότητες των αρχών οι οποίες αξιολογούν και εφαρμόζουν, τις, ελέγχουν τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ε, αλλάζουν και ε, δυστυχώς αναλαμβάνουν αρμοδιότητες οργανισμοί οι οποίοι δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό και δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν σωστά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με μια συγκεκριμένη μορφή αποτυχίας της πολιτικής συνοχής και λυπάμαι που γι' αυτό χρησιμοποιώ το παράδειγμα της χώρας μας. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω την ανάγκη να βρεθεί μια λύση η οποία θα δίδει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να γίνουν οι πραγματικοί δικαιούχοι ενός προγράμματος που τους αφορά. Και αυτό ιδιαίτερα όταν η κεντρική κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι κάποιες επενδύσεις στον τομέα της υγείας, σαν παράδειγμα στην περιφέρεια, είναι απαραίτητες. Ενώ υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε 150 εκατομμύρια για την κατεπίγουσα κατασκευή ενός περιφερειακού νοσοκομείου, η Ρουμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απλά απαραίτητο. Οι τοπικές αρχές λοιπόν έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας, αλλά η κεντρική κυβέρνηση δυστυχώς το απαγορεύει. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τον μηχανισμό μέσα από τον οποίο οι τοπικές αρχές να μπορούν να ολοκληρώνουν τέτοιου είδους υποδομές πέραν της επιθυμίας της κεντρικής κυβέρνησης. Γιατί αλλιώς ε, τα χρήματα τα οποία δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά δεν χρησιμοποιούνται. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές την δυνατότητα να αποκτήσουν ικανότητες και ιδιότητες και νομικού τύπου έτσι ώστε να απορροφούν με μεγαλύτερη ταχύτητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι σαφές ότι σε χώρες όπως τη Ρουμανία υπάρχει μια ένωση ε, των δυτικών περιφερειών. Τέσσερις περιφέρειες έχουν συνεργαστεί σε επίπεδο οργανωτικό και συντονιστικό και προσπαθούν να βρουν λύσεις ε, για την χρηματοδότηση των επιμέρους προγραμμάτων. Εάν δεν ενθαρρύνουμε τέτοιου είδες πολιτικές σε ε, περιφερειακό επίπεδο φοβάμαι ότι θα αποτύχουμε. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε έναν δρόμο 50 χιλιόμετρων και να σταματάμε μέσα στη μέση της υπαίθρου. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η κατασκευή ε, δομών όπως τα νοσοκομεία, οι μονάδες υγείας, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Θα πρέπει λοιπόν οι περιφερειακές αρχές να διαχειρίζονται μόνες τους πλέον ε, τις ε, ευρωπαϊκές πιστώσεις. Μάλετιτς. Να σας ευχαριστήσω να καλωσορίσω για τον Επίτροπο και πολλοί συναδελφοί βίντεο αναφέραν ότι είχαμε την πρότασή σας και ελπίζουμε στον τρομερή διάλογο να υποστηρίξετε και την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, σε ό,τι αφορά τα ανώφια για τη συγχρηματοδότηση. Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο αναφέρθηκε ήδη επίσης ε, η, ο αριθμός των ε, δεκτών απόδοσης από 40-85 ε, ξέρω ότι θέλουμε αποτελέσματα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο να έχει νόημα να γίνεται αυτό με του δείκτες, γιατί θεωρώ ότι ε, περιπλέκει τα πράγματα και σε ό,τι φορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Να ξανασκεφτούμε επίση το θέμα του προγραμματισμού, γιατί το 2018 ήταν το πέμπτο έτος εφαρμογής και νομίζω ότι όλα τα κρατημέλη κατάφεραν να εξαντλήσουν το που κατάφεραν να εξαντλήσουν τα ποσοστά θα είναι ε, αποτελεσματικά και στην εφαρμογή. Έχουμε τώρα και τον κανόνα 5 2. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αποτυπωθεί αυτό και στην ε, εφαρμογή και στην ταχύτητα της όλης διαδικασίας. Ένα άλλο θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι δεν ξεκινήσαμε το παράρτημα 22 και θα πρέπει να συζητήσουμε το γεγονός ότι δεν είναι απόλυτα σαφές πώς θα εκχωρηθούν οι πόροι. Ελπίζω να καταλήξουμε με πιο υψηλά ποσά σε όλες τις διαπραγματεύση για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο και στην πολιτική συνοχή, όπου μειώθηκε το συνολικό ποσό. Τελευταίο θέμα το θέμα ρεσιμότητα, ρεσιμότητας. Ε. Το γεγονός ε, ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση που θα σχετίζεται, ε, όρος που θα σχετίζεται με τη χρηματοδότηση, για παράδειγμα το κρατός δικαίου. Μια καλύτερη λύση θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα οι χώρες που δεν σέβονται το κρατός δικαίου να δίνουν άμεσα στον ευρωπαϊκό προλογισμό ένα 0,2% όπως γινόταν στο 6 pack και στο 2 pack και στο σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Όχι να μπλοκάρονται δηλαδή α, οι χρηματοδοτήσει για του τελικού δικαιούχου, γιατί αυτό δεν αποσκοπεί σε επίπεδο κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν θα μπορούσαμε να το επιδιώξουμε στου τριμερεί διαλόγου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσέλερ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και την κυρία Πίτροπο για την καλή ως τώρα συνεργασία. Όπως και οι προηγούμενοι ομιλητέ, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της διασυνοριακής συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σημείο αυτό να έκανε μια καλή πρόταση σε ό,τι αφορά τα διασυνοριακά προγράμματα και τη διασυνοριακή συνεργασία. Να μην σταματούν όλα αυτά στα σύνορα λοιπόν των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπουν σε ένα καλάθι και να επεκταθούν, να έχουν δυνατότητα επέκτασης μέσω χρηματοδότησης για τις εξωτερικές δράσεις και να φροντίσουμε ότι και πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουμε οι χώρες που έχουν ε, καθεστώς υποψήφιας χώρας ε, ή να μπορούν, ε, για παράδειγμα, να υπάρχει δυνατότητα συνεργασία με τι γειτονικέ χώρε. Ο συνάδελφο από την Ελλάδα επεσήμανε πόσο σημαντικό ήταν το θέμα αυτό ακριβώ τώρα για την Ελλάδα. Το Κοινοβούλιο κατάφερε να πάρει την απόφαση αυτή στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό. Φυσικά θα πρέπει γρήγορα γρήγορα να ξεκινήσουμε τις τριμερεί αντιπραγματεύσει, το τριμερή διάλογο, για να μπορέσουμε εγκαίρως να εγγυηθούμε σωστή πρόσβαση για αυτούς που την επιθυμούν. Γιατί για μένα το θέμα της εθνωριακής συνεργασία αποτελεί θέμα κλειδί πριν, πριν, θέμα στον πυρήνα της πολιτικής συνοχή Γιατί πολλέ χώρε έχουν ε, να πέσουν και πάλι σε εθνικιστικές ιδεολογίες. Ε, γι' αυτό ακριβώς λοιπόν θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή τη διασυνοριακή διάσταση, όπου υπάρχουν λοιπόν ε, αυτές, τα εμπόδια. Ο κανονισμός λοιπόν αυτός αποτελεί μια πολύ σημαντική βάση προς την κατεύθυνση αυτή. Να συγχαρώ επίση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση για ένα καινούριο μηχανισμό για την υπέρβαση των διοικητικών και νομικών εμποδίων σε ό,τι αφορά τη συνοριακή συνεργασία. Αυτό αποτέλεσε ένα πολύ θαραλέο βήμα. Και από όταν ενημερώθηκα σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά και σε κάποιες τοπικές ε, βουλές, Υπήρχε σε πρώτη φάση κάποια αντίδραση και αντίσταση. Εγώ θεωρώ ότι είναι λυπηρό το γεγονό ότι την καταφέραμε εδώ στο Κοινοβούλιο να βάλουμε πιο ισχυρό δεσμευτικό χαρακτήρα για το μηχανισμό αυτό στο Κοινοβούλιο και παραμένει ακόμα αυτός ο θελούσιος χαρακτήρας στην φάση της εφαρμογής. Θα ήθελα να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να επιμείνει παρά την απόφαση αυτή, να προσπαθήσει να πείσει τα κρατη για το πόσο ουσιώδης και ουσιαστικός είναι αυτός ο μηχανισμός μιας και απαλλάσσει από πολλά διοικητικά, γραφειοκρατικά, νομικά εμπόδια, τα οποία έχουν σημασία ιδιαίτερα στις δεσνοριακές περιοχές. Κάθε επιτυχία λοιπόν σας εύχομαι προς την κατεύθυνση αυτή και η Ρουμανική Προεδρία ίσως θα μπορούσε να πείσει τη ρουμανική κυβέρνηση τουλάχιστον να ξεκινήσει το διάλογο τον τρεμερή διάλογο για τα θέματα αυτά τα διασυνοριακά, τουλάχιστον λοιπόν να γίνει τον αρθήριο λάκτισμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις ε, από τα μέλη της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πολλές. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ. Και να σχολιάσετε ενδεχομένω. Ευχαριστώ πολύ και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι σα ακούω γιατί γνωρίζετε σε βάθο την πολιτική αυτή και από εκείνη μπορούμε να βρούμε λύσει. Κατανοώ ότι εργαζόμαστε μαζί, συνεργαζόμαστε εδώ και τέσσερα χρόνια τώρα πλέον. Είναι ο τελευταίος χρόνος λοιπόν που θα έχουμε και ίσως θα μαζί σας πάλι στο τέλος του έτους για να προσπαθήσω να απαντήσω όμως τώρα στις ερωτήσεις σας, στα σχόλιά σας. Για την κυρία Κωνσταντσε Κρέλ. Ξέρετε πολύ καλά ότι η πολιτική αυτή αποτελεί έναν από τους πυλώνες της πολιτικής μας. Σας ευχαριστήσω πολύ για την υποστηρίξή σας και για την υποστηρίξη για τις προτάσεις απλοποίησης. Γιατί προφανώς εκτιμούμε ιδιαίτερα τη βοήθειά σας. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην επανέλθουμε στους ίδιους κανόνες. Που κάνουν όλο τον κόσμο να παραπονιέται. σε όλες τις χώρες υπάρχουν παράπονα για την γραφειοκρατία, για το πόσο ε, πολύπλοκα είναι τα συστήματα. Έμα ε, νομίζω μετά από 25 χρόνια με τους ίδιους κανόνες έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να γίνει ε, μια μαζική απλοποίηση. Για τον προπολογισμό καθε αυτό χαίρομαι που καταφέραμε να πετύχουμε το πιο ψηλό φάκελο για την πολιτική συνοχή σε 73 δις για τις 27 χώρες αλλά φυσικά θα προτιμούσα να ήταν πιο υψηλή πρόταση για τον προπολογισμό για τη δική μας πολιτική. Δεδομένων όμως των ε, δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε, ξέρετε ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα και να πετύχουμε έναν ε, φιλόδοξο προπολογισμό. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην σοφία του θα εκχωρήσει πιο πολλούς πόρους στην πολιτική μας. Ας ελπίσουμε. Ας ελπίσουμε και ας υπολογίζουμε στην γενεδορία του Συμβουλίου. Για τους σημερινούς διαλόγους ελπίζουμε να ξεκινήσουν άμεσα μετά από την έγκριση της Ολομέλειας σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη διαχείριση των προγραμμάτων. Είναι σημαντικό θεωρώ αυτό το σκέλος για την απλοποίηση. Η κυρία Τόμασιτς, 80% των ε, πόρων μας θα περάσει στην επόμενη προγραμματική περίοδο σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Και εδώ πιστεύω ότι η απλοποίηση και η επικοινωνία είναι σημαντικά ζητήματα. Το θέμα δεν είναι μόνο τα χρήματα. Έχουμε πολλά προγράμματα, πολλά εργαλεία και ξέρουμε ότι η πρώτη απόφαση που έλαβα όταν ε, ξεκίνησα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αυτή η Task Force για την καλύτερη εφαρμογή σε οκτώ κράτη-μέλη που υστερούσαν. Πραγματικά τα βοηθήσαμε. Ήταν ικανοποιημένοι. Και όλοι οι εμπειρογνώμονες βοήθησαν τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές, ε, έδωσαν συμβουλές και όντως τα νεα κρατημέλη έχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τις ε, διοικητικές ε, ικανότητες τους. Εγώ είμαι μεγάλη υπερμαχός αυτής της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των χωρών που χρησιμοποιούν τέτοιου πόρου. Και αντίδρα σε ό,τι αφορά παλιέ και νέε χώρε, όπω είναι η Κροατία. Είναι σαφές ότι τα νέα κράτη-μέλη που προστάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια το 2004 έχουν σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο στα ευρωπαϊκά ταμεία. Έχουμε χώρε όπω η Βουλγαρία που 80% όλων των δημόσιων επενδύσεων γίνονται με ευρωπαϊκού πόρου και στη Ρουμανία 60% των δημοσίων επενδύσεων. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να παρέχουμε υποστήριξη να συνοδέψουμε όλα τα κράτη-μέλη στις διαπραγματεύσεις στη νέα προγραμματική περίοδο και σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες για τη νέα προγραμματική περίοδο. Αλλά να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε εκεί και στην προγραμματική αυτή περίοδο αυτή. Τον κύριο Φαμίλτεμπριχ να ευχαριστήσω για τα σχόλιά του. Είπατε σωστά ότι η ποιότητα των προγραμμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήθελα να πω ότι οι πληρωμέ τελευταία στιγμή είναι κάτι το είναι, που είναι πολύ κοινό. Όχι μόνο στη Ρουμανία. Πολλέ χώρε έχουν υποβάλει το Δεκέμβριο τέτοιε πληρωμέ. Τώρα φυσικά είναι καθήκον των ελεκτών να ελέγξουν την ποιότητα των προγραμμάτων αυτών. Και όντω, στην περίπτωση τη Ρουμανία, Στην αρχή του 2018 είχαμε κίνδυνο αποδέσμευσης από τα περιφερειακά ε, προγράμματα πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ και αλλάξαμε λειτουργικά προγράμματα προκειμένου να μεταφέρουμε πόρους από τομείς χαμηλής απορρόφησης ε, όπως ε, στις μεταφορές σε άλλους τομείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις το καλύτερο πρόγραμμα στη Ρουμανία, το πιο επιτυχέ. για την υγεία, για παράδειγμα. επίση εναλλακτικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα αυτά των ασθενοφόρων, ένα πρόγραμμα το οποίο υποτίθεται θα το χρηματοδοτούσαμε σε εθνικό επίπεδο, με εθνικού πόρους, αλλά κατόπιν αιτήματο τη ρουμανική κυβέρνηση, συμπεριλήφθησε στα ευρωπαϊκά ταμεία. Όπως σα είπα λοιπόν υπήρχε αυτό το στοιχείο ευελιξίας για όλα τα κράτη-μέλη για την αλλαγή τέτοιων λειτουργικών προγραμμάτων σε ό,τι αφορά πολλά προγράμματα, τους μετανάστες και το καθεξής. Και ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να μην χάνουν λεφτά. Να σας διαβεβαιώσω όμω ότι ακολουθούμε του κανόνε. ανεξάρτητα από το κράτος μέλος το οποίο μιλάμε και κάνουμε εξίσου αυστηρούς ελέγχους σε όλα τα κράτη-μέλη. Χωρίς να διστάζουμε. Όντως, δεν είχαμε ούτε πόρους, ούτε χρήματα για να ξεκινήσουμε τέτοιο έλεγχο των προγραμμάτων. αλλά οι ελεκτές ελέγχουν πλέον το κατά πόσο είναι νόμιμα τα προγράμματα ή όχι. Είναι σημαντικό όμως ότι αποφύγαμε αυτή την αυτόματη αποδέσμευση. Πλέον λοιπόν καλύπτονται τα χρήματα από τα προγράμματα και τα αιτήματα πληρωμών, αλλά θα δούμε κατά πόσο θα είναι ποιοτικά ή όχι. Όπως και να έχει ισχύουν για όλες τις χώρες ε, οι ίδιοι κανόνες. Κύριε Παπαδημούλη, σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Συναντήθηκα με τον Υπουργό για τα θέματα τα ψηφιακά, πολύ σημαντικό θέμα για την Ήπεθρο. Και φυσικά και ελπίζω ότι θα πετύχουμε το συντομότερο δυνατόν μια συμφωνία, να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο. Είμαστε έτοιμοι και από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς είσαστε έτοιμοι. Και ελπίζω ότι και το Συμβούλιο θα είναι έτοιμο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και αύριο ακόμα για τα θέματα της δυσνοριακής συνεργασίας. ανυπομονούμε. Μου φαίνεται ότι τα πράγματα καθυστερούν στο Συμβούλιο, γιατί βλέπω ότι και εσείς είσαστε έτοιμοι και πρόθυμοι. Ελπίζω λοιπόν να ξεκινήσουμε τους ε, τριμερείς διαλόγους για το θέμα της ε, Πουγουδμούδου. Υπήρχε η διαφωνία για το όνομα, μιας και κινούμαστε τώρα προς τη σωστή κατεύθυνση από ό,τι φαίνεται. Φυσικά τα πράγματα θα διευκολυνθούν μόλις ξεκινήσουν να ισχύουν οι λειτουργικοί κανόνες μεταξύ των ε, δύο χωρών. Για το θέμα των ε, νησιών. Είναι μια ερώτηση αρκετά κοινή, συνηθισμένη από τον κύριο Παπαδημούλη και την κυρία Μπρέσο. Ξέρετε ότι προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις συγκεκριμένε ανάγκες των περιεχών και όλες οι εκθέσεις και αναφορές καταδεικνύουν ότι υπάρχει Μεγάλη, υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις σε πολλές ε, περιοχές της Ευρώπης. Ε, έχουμε κάνει και συζήτηση και στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι στη νέα πρόταση τα κρατη έχουν επιφέρει ευελιξία σε ό,τι αφορά την εκχώρηση των πόρων ε, στο ιστορικό των χωρών. Στα κρατη λοιπόν επαφήνεται να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις ε, συμφωνίες αυτές για τις ανάγκες των περιφερειών. Θα θέλαμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο να υπάρχει πιο α, υποστήριξη μέσω των εργαλείων περιφερειακής ε, και ταφικής ε, ενοποίησης. Θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε αυτό και στο μέλλον. Για την απλοποίηση όμως και προκειμένου να υπάρχει απλοποίηση, δεν έχουμε ακόμα επεξεργαστεί το πεδίο εφαρμογή και νομίζω ότι σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να αποφασιστεί αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις απόκτρες περιοχές και τις περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και εδώ υπάρχουν ε, συγκεκριμένες εκχωρήσεις. για την εκχώρηση πόρων. Ξέρετε πολύ καλά ότι χρησιμοποιούμε το ΑΕΠΑΝΑ κατά κεφαλή. Η μέθοδος Βαρολίνου, όπως ε, αποκαλείται, είχαμε πάνω από 20 σενάρια και διαπιστώσαμε ότι αυτό ήταν το πιο ενδεδειγμένο και το πιο ισορροπημένο ως μέθοδος. Η μέθοδος αυτής αρχικά είχε χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία φακέλων, εθνικών φακέλων για την περίοδο μετά το 2000-2006 είναι μια μέθοδος που βασίζεται στην ε, περιφερειακή και τοπική ευμερία. Είναι ποσοστό του κατακεφαλήν ΑΕΠ και βάλαμε και κάποιους επιπλέον ε, δείκτες όπως ε, αλλαγή κλίματος, ανεργία των νέων, μετανάστευση και το καθεξής. Και έγινε μια προσαρμογή. Άρα από πλευράς μας και με το δίκτυο ασφαλείας που είναι σημαντικό και αυτό πιστεύω γιατί πολλά μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο και θα είχαν χάσει πολύ πιο πολλά σε σχέση με την πρότασή μας. Άρα θεωρώ ότι είναι ισορροπημένη τελικά η πρόταση. Όπως και να έχει. Ξέρετε πολύ καλά ότι στο τέλος των διαπραγματεύσεων τα πράγματα πάντα δυσκολεύουν και περιπλέκονται. Χρειάζεται και χρόνος για να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Αλλά διάφοροι Συζητήσατε να διευκρινίσουμε το χρονοδιάγραμμα. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι είναι ανθρωπίνο δυνατό στη φετή αυτή. Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί το επόμενο κοινοβούλιο. Πότε θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, πότε θα είναι λειτουργικό. Και εγώ ανησυχώ για την ε, τελευταία έγκριση του Πουδουπού. Θα πρέπει να δε αποδείξουμε ότι κάτι μάθαμε και από τα παθήματα του παρελθόντος. Γιατί σε πολλά κρατημέλη υπήρχε καθυστερημένη έγκριση λόγω καθυστερημένης έγκρισης του, των κανονισμών. Και ο πρόεδρος Γιούγκερ και πολλοί άλλοι το Δεκέμβριο είπαν ότι θα πρέπει μέχρι τις ευρωεκλογές να έχουμε πετύχει τη συμφωνία για το Πουδουπού Μέχρι το φθινόπωρο του 2019 πλέον είναι η ημερομηνία αυτή και φυσικά είμαι αισιόδοξη ότι θα το πετύχουμε αυτό. Για την ανάπτυξη της υπέτρου. Ο κύριος Νομποκόφ αλλά έφυγε. Φυσικά και σέβομαι την πρότασή του, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβα, υπέβαλε την πρότασή της και θα δούμε ποια θα είναι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στο τριμερή διάλογο για τα ποσοστά σε χρηματοδότηση τώρα. Κυρία Μάλατιτς. Νομίζω ότι θα συμπεριληφθεί στι διαπραγματεύσει. Ο καλύτερο τρόπος είναι να ξεκινήσουμε το συντομότερο των της διαπραγματεύσει και μετά βλέπουμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Η πρότασή μας για τη χρηματοδότηση είναι να δοθεί μεγαλύτερη υπευθυνότητα στα κράτη-μέλη και το κράτος δικαίου για τον ε, ευρωπαϊκό υπολογισμό είναι όρος και σημαντικός ε, για τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό να αναλάβουμε τις ευθύνε τους. Να δούμε τώρα φυσικά γιατί θα εγκρίνετε τις δικές σας προτάσεις, θα δούμε και ποια θα είναι η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου και τι μηχανισμός τελικά θα επικρατήσει. Κύριε Μπουτά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσέγγισή σας και θα ήθελα να πω ότι για μένα είναι σημαντικό να βοηθούσουμε τα κράτη-μέλη, αλλά εκ παραλλήλου δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τίποτε αναφέρατε τα τρία περιφερειακά νοσοκομεία. Αυτό επαφείται στο Υπουργείο Υγείας. Ξέρω ότι υπάρχει αυτό το αίτημα, αλλά χρειάζεται αίτημα από τις εθνικές αρχές για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Φυσικά έχουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Και υποχρέωση να εκχωρούνται 6% των πόρων στις τοπικές αρχές άμεσα, από τις τοπικές αρχές άμεσα. Ακόμα και για την τρέχουσα πραγματική περίοδο. Έχουμε τα ευρωπαϊκά ταμεία τα οποία τα είναι υπό διαχείριση από τις Δήμους άμεσα. Είναι σημαντικό αυτό το γεγονός λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η τοπική στρατηγική ανάπτυξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον σωστό προγραμματισμό και την απόδοση των μέτρων και τις δράσεις που θα αναλάβουμε. Έχει σημασία αυτό, γιατί δεν μπορούμε εμείς στις Βρυξέλλες να γνωρίζουμε καλύτερα ε, το πού και πώς θα επενδύσουμε. Αλλά μερικές φορές και οι εθνικές αρχές είναι αυτές που δεν είναι τόσο ενημερωμένες όσο οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την υπομονή σας, σας εξάντλησα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν το ταχύτερο δυνατόν να ξεκινήσουμε τις τριμερείς διαπραγματεύσεις. Η συνεργασία μαζί σας είναι κάτι το οποίο περιμένω με πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία. Θα έπρεπε να έχουμε ήδη ξεκινήσει. Ας μην αναβάλουμε λοιπόν, ας προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν και είναι σαφής ο ρόλος σας ως συνεισηγητές και συνομοθέτες. Σας ευχαριστώ Επίτροπε. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε τη Ρουμανική Προεδρία σήμερα. Θέσαμε όλες τις ερωτήσεις που έπρεπε και θέλουμε να μην καθυστερήσουν οι διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ για όλες τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία μαζί σας και ελπίζω να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις το ταχύτερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, αυτό ήταν το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διατάξεώς μας για σήμερα. Είχαμε πάρα πολλή δουλειά μέχρι σήμερα. Πήρατε και ένα mail με τις αποφάσεις των συντονιστών. Μπορούμε να τις εγκρίνουμε παρακαλώ. Ευχαριστώ, δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στα διάφορα. Θα ήθελα μία παρατήρηση μόνο να κάνω, ότι σήμερα, όπως θυμίστε, είχαμε προγραμματίσει να πιούμε κάτι μαζί για να πάει καλά η χρονιά. Τα ποτά θα τα βρούμε στον χώρο Ι, ε, ε δηλαδή, στον πρώτο όροφο, στις 6. Ό,τι πρέπει δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχω άλλο ένα μήνυμα. Η συνάντησή μας η επόμενη στις 14 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. 14 Φεβρουαρίου επαναλαμβάνω στο Στρασβούργο. Ακυρώθηκε η συνεδρίαση της 7 η Φεβρουαρίου και θα συναντηθούμε στις 14 στο Στρασβούργο. Ευχαριστούμε την επιμελητία λέει η Πρόεδρος και όλους όσους πήρατε μέρος στη συνάντηση.